Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons commencer. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρία ανταλλαγής απόψεων με τον ε, υποψήφιο επίτροπο κύριο Καρλ Ντεγκούχτ προς διευκόλυνση της κατανόησης όλων. Θα συνεχίσω. Στα αγγλικά λέει η πρόεδρος. I would like to ήθελα επισήμω να κηρύξω την έναρξη τη ανταλλαγή των απόψεων και για λογαριασμό τη Επιτροπή Ανάπτυξη να καλωσορίσουμε θερμά τον Κάρελ Ντεχιούχτ, που είναι ο υποψήφιο Επίτροπο για Ανθρωπιστική Βοήθεια και Ανάπτυξη. Επί 15 χρόνια διατέλεσε μέλο του Κοινοβουλίου. Έχουμε μία ώρα και 45 λεπτά για να δουλέψουμε σκληρά. Και για αυτό θα Περίωσα αυτή την εισαγωγή στο να σας εξηγήσω την διαδικασία πριν αρχίσουμε την ανταλλαγή των απόψεων. Ο προηγούμενο επίτροπο αυτού του χαρτοφυλακίου Λουί Μισελ παραιτήθη από μέλη τη Επιτροπή και γι' αυτό το λόγο είμαστε εμεί οι αρμόδιοι να οργανώσουμε αυτή την ανταλλαγή των ε, απόψεων με τον υποψήφιο επίτροπο Καρλίτε Χίχτ. Και έχουμε την προσωπία από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, οι οποίε θα συμμετάσχουν σε αυτή την ανταλλαγή των απόψεων. Ο βασικό του σκοπό αυτή τη συνέντευξη των απόψεων είναι να προετοιμάσουμε την ε, έγκριση ε, του ορισμού ή διορισμού αυτού του επιτρόπου εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέραν αυτών τώρα, αυτή η διορισμου αυτου του επιτροπου εκ μερου του ευρωπαικου κοινοβουλιου τωρα αυτη η ανταλλαγη των απόψεων πρόκειται να δώσει στην ε, Επιτροπή μα την ευκαιρία του να τον γνωρίσουμε καλύτερα. γνωρίζουμε, για να γνωρίσουμε του του, να, να δούμε τι εμπειρία έχει και σε περίπτωση που εγκριθεί η υποψηφιότητά του, με αυτή την ανταλλαγή των απόψεων θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια σχέση συνεργασία από τώρα ε, και εμεί ω Επιτροπή με τον υποψήφιο Επίτροπο. Και τελευταίο, αλλά σημαντικό, με την ανταλλαγή των απόψεων θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση για την εργασία και το έργο του Επιτρόπου ε, στη συνέχεια ε, συγκρίνοντας, αντιπαραβάλλοντας το, το έργο του με τις δηλώσει του και τα σχέδια που θα εξαγγείλει. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, σας υπενθυμίζω. Για άλλη μια φορά, τι προβλέπετε. Η ακρόαση θα κρατήσει μία ώρα και 15 λεπτά. Πρώτα-πρώτα θα έχουμε μια, ένα αρχικό γύρο δηλώσεων εκ μέρους των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή μας όσον αφορά τις προτεραιότητες τους για τον τομέα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό θα κρατήσει 9 λεπτά. Κατά δεύτερον, θα ακούσουμε για 15 λεπτά τι έχει να μας πει ο υποψήφιος. Κατόπιν θα έχουμε 9 γύρους ερωτήσεων και απαντήσεων. Ε, πολιτική ομάδα, 4-5 ερωτήσεις. Ε, ε, μισό λεπτό ή 45 δευτερόλεπτα για τα σχετικά ζητήματα βέβαια και κατόπιν θα απαντά ο υποψήφιος επίτροπος ε, επί 5 λεπτό ή 6 Στον τρίτο γύρο οι συνάδελφοι της ε, ΑΦΕΤ μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και για τον έκτο γύρο τα, τα, τα, τα μέλη της Επιτροπής των, του Εξωτερικού Εμπορίου μπορούν να υποβάλουν ε, τις δικές ερωτήσεις και κατόπιν Έχουμε άλλα τέσσερα λεπτά. Η κάθε επιτροπή αυτέ τι ερωταπαντήσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, ούτω ώστε να μπορέσουμε να με δίκαιο τρόπο να δώσουμε ευκαιρία σε όλους να υποβάλουν ερωτήσει ή στον υποψήφιο ε, επίτροπο. Και σας ε, προειδοποιώ, αν υπερβεί τα χρονικά όρια, θα ε, σα αφαιρέσω τον λόγο και θα λάβει τον λόγο ο επόμενο συνάδελφο. Ο υποψήφιο στι 5 η ώρα θα κλείσει την συνεδρίαση με κάποιε καταγγελικέ παρατηρήσει και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι δικέ μου. Θα βάλουμε τα αποτελέσματα αυτά τη συζήτηση ε, στου πρόεδρου των Επιτροπών και των Πρόεδρων Κοινοβουλίου ε, με τη μορφή μια επιστολή. Οι δε συντονιστέ τη Επιτροπή ε, τη Ανάπτυξη πρόκειται στι 3 Σεπτεμβρίου να συναντηθούν εκτάκτω, ώστε να αναλύσουν τα όσα έγιναν και 14 με 17 Σεπτεμβρίου που έχουμε την Ολομέλεια στο Στρασβούργο πρόκειται επισήμως να γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή. Ο πρώτος γύρος τώρα. Θα ακούσουμε τις ε, δηλώσεις, τοποθετήσει των πολιτικών ομάδων της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου. Θα ακούσουμε τι προτεραιότητες έχουν όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια οι πολιτικές ομάδες. Η Μίτσελ του Ευρωπαϊκού Λεγόματος έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κερδίζουμε την παρουσία του υποψηφίου επιτρόπου. Ελπίζουμε να έχουμε δημιουργική συνεργασία και βλέπουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες διπλά τιμωρούνται ε, για την οικονομική κρίση. Το 0,7% αυτή η συμβολή του ΑΕΠ που τα κράτη-μέλη είπαν ότι θα δώσουν είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Μια που υπάρχει αυτή η κρίση επομένω. Αυτή η κρίση φέρνει συρρήκνωση του ΑΕΠ. Οπότε και αυτή η συμβολή φυσικά και μειώνεται σαν ποσό. Αλλά ε, δεν συγκρώνεται το, το ποσοστό. Επομένω τα κράτη δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρηθεί αυτό το 0,7%. Στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι η αμυντική συνεργασία θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε δράσεις ε, ειρήνη, ελευθερίας, δικαιοσύνη, να βοηθήσουμε την παραγωγικότητα, να βοηθήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα στι ανεπτυσσόμενε χώρε. Εσεί τι λέτε, υποψήφια επιτροπή. Αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ε, βιωτικό επίπεδο, διαφάνεια, καλή διακυβέρνηση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε το επιχειρηματικό πνεύμα και να γίνει κάποιο είδους αναδασμός ει όφελος των ακτιμών. Και έτσι να χτυπήσουμε τη φτώχεια. Παρακαλούμε αυτό, και υποψήφιο επίτροπε, να καταστεί προτεραιότητά σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Έχει απόλυτο δίκιο Γκέι Μίτσελ όταν λέει ότι το 0,7% είναι το ελάχιστον το οποίο θα πρέπει εμείς να ζητούμε και να πρεσβεύουμε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να φροντίσει ο Κάλ Ντεχέχτου τους επόμενους μήνες στα κράτη-μέλη αν μη τι άλλο να τηρήσουν αυτή την υπόσχεση και όχι προς τα κάτω, προς τα πάνω. Ένα αυτό. Μετά η κρίση, η ε, χρηματοοικονομική και επιστοτική, πώ θα τη, τη θα και πώ θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για αναπτυγμένα κράτη. Το ίδιο ισχύει για την κλιματική ε, κρίση ε, τους τελευταίους μήνες ήταν πρωτοσέλιδο αλλά έχει επισκιαστεί. Ε, υπάρχουν κάποια μέτρα απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Πού είναι η χρηματοδότηση στα αναπτυσσόμενα κράτη. Δεν έχει εξασφαλιστεί σε κανένα βαθμό. Εσείς τι θα κάνετε, ρωτάει η σοσιαλδημοκρατική ομάδα, γιατί είναι προτεραιότητα για μας. Τρίτον, η συνοχή και η συνέπεια στην πολιτική μας. Ξέρει η πρόεδρος κυρία Παζολή ότι επίκειται μια ε, συμφωνία αλλιευτική με τη Γουινέα, όπου διαφυλάσσονται τα δικά μας συμφέροντα, των αλλιών μας δηλαδή, αλλά όχι των αλλιών της Γουινέας και ακόμα λιγότερο του περιβάλλοντος της. Τι γίνεται εκεί. Ελπίζω να αφιερώσετε και εκεί ενέργεια. Και ένα τελευταίο. Ελπίζω κάποια στιγμή, ίνσαλα, πρώτα ο Θεός να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και να έχουμε και Ευρωπαίο Επίτροπο για αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι εσείς φιλοδοξείτε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά λέτε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να αποσασιοποιηθεί ε, ε, από την εξωτερική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Πώς το βλέπετε. Βεβαίως συνδέονται η εξωτερική πολιτική και η αναπτυξιακή, αλλά η αναπτυξιακή ε, πολιτική κυρίως στρέφεται ε, στο συμφέρον της ανάπτυξης, των φτωχών κρατών δηλαδή και όχι το συμφέρον ή τα συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτά έχει κατά κύριο λόγο υπόψη της εξωτερική πολιτική. Εκεί υπάρχει ένα θέμα συνέχειας και συνοχής. Για να είναι κάποιο ανεξάρτητος θα πρέπει λοιπόν να είναι ανεξάρτητα θεσμικά όργανα και ανεξάρτητη γενική διεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, <clears throat> Mr. Berman. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέρμαν, ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ο κύριος Δεκίχτ Θα αναλάβει τη θέση αυτή μετά τον κύριο Λουί Θα τον διαδεχτεί. Και εγώ θα ήθελα να αποτίσω φοροτιμή στο έργο του κ. Μισελ ω Επιτρόπου τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό που περιμένουμε από τον μελλοντικό Επίτροπο. Ναι, νομίζω ότι μπορείτε να χειροκροτήσετε. Τα αξίζει τα χειροκροτήματα ο κ. Μισελ. Αυτό που προσδοκούμε λοιπόν από τον ε, μελλοντικό Επίτροπο είναι αυτό που περιμένουμε από κάθε παράγοντα στην ανάπτυξη. Συνοχή στην προσέγγιση, συμπληρωματικότητα των δράσεων και καλείστε να καλύψετε δύο σημαντικούς τομείς στην υπηρεσία σας, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, ανάπτυξη αυτή καθεαυτή από την άλλη. Ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια, ανέκαθεν, είναι μια απάντηση στις διάφορες ανεπάρκειες και αποτυχίες μας. Η αναπτυξική βοήθεια είναι το σκέλος των αρμοδιοτήτων σας, που είναι λιγότερο θεαματικό, περισσότερο, λιγότερο θα περάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις τηλεοράσεις, αλλά θα πρέπει εκείνη να εκτυπώσετε όλοι σας την δεξιοτεχνία. Υπάρχει λοιπόν μια επιτροπή, ένας ε, επίτροπος με ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες και 27 κράτη-μέλη. 28 λοιπόν ε, συμμετέχονται στην όλη διαδικασία τη αναπτυξιακή βοήθειας. Ελπίζω ότι θα έχετε όλη την απαραίτητη στήριξη για να φέρετε με επιτυχίες πέρα στα καθήκοντά σα. Τα οποία πλαισιώνονται από την δήλωση των Παρισιών, τη συμφωνία τη Κοτονού και την μερική σύναψη των συμφωνιών οικονομικής εταιρική σχέσης. Βλέπουμε τι γίνεται και με τις κλιματικές αλλαγές ταυτόχρονα. Αυτό που περιμένουμε από εσάς λοιπόν κύριε Τεκόφτ είναι σε σχέση με όλους τους απεσιόδοξους που σχεδιάζουν μια θλιβερή εικόνα για την ανάπτυξη, να δράξετε την ευκαιρία εσείς, η Επιτροπή σας και η Γενική σας Διεύθυνση, ώστε να δώσετε έμφαση στην πραγματική έννοια, την ουσία της ανάπτυξης. Ο κύριο Στάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα ε, τον Κάρλ Ντεχιόχτ εδώ. Καλωσορίσατε και πάλι. Έρχεστε εδώ, κύριε Ντεχιόχτ, ε, ενώπιον βουλευτών που με πάθος ε, εργάζονται στην αναπτυξιακή συνεργασία για τα δικαιώματα, την ευημερία ε, των φτωχοτέρων που πλήττονται περισσότερες χώρες αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η εντολή σας αυτή για ανθρωπιστικά ε, και άλλα χαρτοφυλάκια είναι απλώς ένα σκαλοπάτι, ένα εφαλτήριο για να πάτε σε άλλη θέση επιτρόπου που τη θεωρείτε σημαντικότερη. Και αν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν καταβάλλετε προσπάθειες να μας στείλουν ε, ε, κάποιον άλλο, ή να διατηρήσετε αυτό το χαρτοφυλάκιο αν το θεωρείτε εσείς σημαντικό. Οι δικές μας προτεραιότητες είναι εξής, θα επανέλθουν οι συνάδελφοί μου. Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα για τις συμφωνίες εταιρική σχέσης και οικονομικές ε, αυτές γίνονται από θέση ισχύω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό δεν βοηθάει τους στοχοτέρους στις χώρες αυτές τι πιστεύετε γι' αυτό. Δεύτερον, επίκειται η σημαντική διάσκεψη Κοπενχάγη για το κλίμα. Το κλίμα και η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και είναι σαφές ότι η κλιματική αλλαγή ε, προκαλεί πάρα πολλά θύματα. 300.000 νεκρού ακούω 325 εκατομμύρια απειλούνται ε, με προσφυγιά πολλές φορές ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τι θα κάνετε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες εν ώψη λοιπόν αυτή της σημαντική συνόδου κορυφής τέλος Οκτωβρίου. Και τέλος η χρηματοπιστωτική κρίση και πάλι δυσανάλογα πλήττει τις φτωχέ χώρες. Εσείς τι θα κάνετε, τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε τα μέσα που ε, έχουμε στη διάθεσή μας και τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας να υλοποιούνται. Τέλος, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Δίβα έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τεχόρτ έρχεται σε μια πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή για το χώρο της αναπτυξιακής βοήθειας και της ανάπτυξης και θα υποφεληθεί από το σκληρό έργο του προηγούμενου επιτρόπου, του κ. Λεμισέλ, που βρίσκεται μαζί μας και τον χειροκροτώ και εγώ, τον επικροτώ μάλλον για, το, για τις προσπάθειες που έκανε για να φέρει πέρασμα επιτυχία το έργο του. Οι συντηρητικέ και μεταρρυθμιστικέ προτεραιότητε του Κοινοβουλίου θα επικεντρωθούν στι λύσει που επεξεργαστήκαμε με το ΕΛΚ στο προηγούμενο θητεία του Κοινοβουλίου. Η πρώτη μα προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε αυτέ τι προτεραιότητε προκειμένου να καταπολεμήσουμε την ένδια και να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για το χρήμα των φερολογουμένων μα. Η κατευθυντήρια γραμμή μα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανθρωπίνη εξωπρέπεια κάθε ανθρώπινου όντω στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Να Προσθέσω τρει αποχρώσει εδώ. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται ουδέτερη ε, αναπτυξιακή βοήθεια για να υπάρξει σταθερότητα και πρέπει να αποφύγουμε τις ευλογικές επιδοτήσεις και τους εμπορικούς φραγμούς που έχουν βλάψει τόσο πολύ. Έπειτα, οικοδόμηση δυνατοτήτων με την, ε, με την, ε, την έβνοια της ε, απασχόλησης είναι κάτι που μόνο μέσω κοινωνικών υπηρεσιών και τη συμμετοχή των κοινωνία των πολιτών μπορεί να επιτευχθεί. Με θεσμού σταθερού με θέση των τιμών που να μην βασίζεται σε εμπορικό κόσμο τη απορρίθμιση. Θα πρέπει να προωθήσουμε και να ευνοήσουμε την καλή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη των δεξιτεχνών των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μια ανεξάρτητη θέση στην ε, διεθνή αγορά. Και επίση η αποστράγγιση εγκεφάλων ε, από τι αναπτυσσόμενε χώρε είναι ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο. Διότι οι αναπτυσσόμενε χώρε δεν μπορούν να χάσουν κι άλλου ε, αξιόλογου ανθρώπου του. Πρέπει να δούμε τα φαινόμενα τη κυκλική μετανάστευση λοιπόν ω προ αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την αρχική μου παρέμβαση. Ευχαριστούμε κύριε Ντέβα. Η κυρία Γκαμπρίελε Τσίμερ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Γενικά χρειάζεται ένας νέος προσανατολισμός των σχέσεων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προς χώρες του Νότου. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια μπορεί να ανήκουν ε, στους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής, συγγνώμη, αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά ταυτόχρονα ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα παγκόσμια προβλήματα και για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Γι' αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, τι πιστεύετε, ακόμα και είναι μεταβατικό αυτό το πόστο που αναλαμβάνετε και ε, θα με ενδιαφέρε λοιπόν πώς αξιολογείται τη μέχρι τώρα πορεία μας ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια, ποια θα πρέπει να είναι η αναπτυξιακή πολιτική, ποια είναι η σχέση των χωρών του Νότου με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην είναι δωρητές και ε, δικαιούχοι, αλλά να είναι ισότιμοι σε μια εταιρική σχέση, όχι μια σχέση εξουσίας. Ε, και τι γίνεται με τους πόρους που έχουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για να υλοποιηθούν οι στόχοι της χιλιετίας. Και τι θα κάνετε για να ακουστεί περισσότερο ε, η φωνή της Αφρικής. Στους G20 κάποια στιγμή θα εμφανιστεί η Αφρική, να μην αποφασίζουν ε, οι μεγάλοι της γης ε, ε, ρήμην της Αφρικής. Uh, Ευχαριστούμε. Και τώρα, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Για ένα τέταρτο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη χαρά για μένα η ευκαιρία που έχω σήμερα να απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Επίτροπος για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, ε, διατέλεσα 14 χρόνια ευρωβουλευτής. Κανένας δεν μπορεί περισσότερο από μένα να αξιολογήσει και να εκτιμήσει το ουσιώδη ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, το να γίνει η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο δημοκρατική και πιο υπόλογη. Σήμερα έχω την περηφάνεια να πω ότι και προσωπικά συνεισέφερα στην ενίσχυση των ελεκτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βοηθήσω στο να διαμορφωθεί αυτό που σήμερα είναι γνωστό στη διαδικασία ακρόαση, όπου ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί και εκτιμά τη γενική ικανότητα, την ευρωπαϊκή προσήλωση και την προσωπική ανεξαρτησία των υποψηφίων επιτρόπων ε, πριν ε, ψηφίσει για να εγκρίνει ένα νέο σύνολο επιτρόπων. Από την πρώτη αυτή μου εμπειρία ως Ευρωβουλευτής μετακόμισα στο Συμβούλιο ως υπουργό ενός κράτους μέλους και σήμερα ελπίζω να ε, τετραγωνίσω τον κύκλο της Ευρωπαϊκής μου σταδιοδρομίας ως Επίτροπος και να δεχθώ την υποστήριξή σας για το πρόγραμμά μου. Για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας τη Επιτροπής, ο πρόεδρος Μπαρός αποφάσισε να μου αναθέσει το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Λουί Μισελ, που είναι τώρα Ευρωβουλευτής ή συνάδελφός σα, και στον οποίο θα ήθελα να αποτίσω ένα φόρο τιμής για τη γερή και καλή δουλειά που έκανε στην ευρωπαϊκή ε, πολιτική ε, συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Και ε, βοήθησε να βαθυνθούν οι σχέσεις μας με τις χώρες ΑΚΕ. Σε κάποιο βαθμό η προεργασία του αυτή μου διευκολύνει σήμερα το δικό μου έργο, καθώς κληρονομώ ένα πλαίσιο πολιτικής και συνενετικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους επόμενους μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απομένει, ιδιαίτερα σε περιόδους παγκόσμιας ύφεσης. Εδώ δεν μπορώ παρά να συμμεριστώ τους στόχους που μέχρι τώρα έχουν εμπνεύσει αυτές τις πολιτικές και είμαι πλήρως ε, στρατευμένος στην υπόθεση αυτή να συνεχίσω την εφαρμογή τους επόμενους μήνες. Επιπλέον δε, πράττοντας ε, ούτως, δεν πρόκειται να προεξοφλήσω ούτε να δεσμεύσω μακροπρόθεσμα οποιασδήποτε άλλε αλλαγέ και επιλογέ θελήσει να κάνει ο επόμενο επίτροπο και διάδοχό μου. Δεχόμενο αυτό το πόστο, θεωρώ ότι έχω και τα απαραίτητα και τα σωστά διαπιστευτήρια να συνεχίσω τη δουλειά με τρόπο ε, αξιοπιστό και επαγγελματικό προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εξωτερική προβολή από την ε, ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική ανάπτυξη. Ως Ευρωβουλευτή συμμετείχα ενεργά στην τότε Συμβουλευτική Συνέλευση ε, ΑΚΕΟΚ, που τώρα είναι η ε, Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ως Βέλγος Υπουργό Εξωτερικών, είχα εμπειρία που με βοήθησε πολύ ε, πρόσφατα σε πολλά θέματα που σήμερα είναι στην καρδιά της διεθνούς συνεργασίας και κρίσιμα για τις σχέσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσομένων κρατών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επίκυνται σημαντικά ζητήματα και προθεσμίες. Και πρώτα απ' όλα η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, αυτή πλήττει σήμερα τις αναπτυσσόμενες χώρες που είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθούμε, διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει ε, περαιτέρω ε, πολιτική και κοινωνική αστάθεια στον κόσμο. Σε τρει εβδομάδε, σε διεθνέ επίπεδο, η Σύνοδο των G20 στο Πίτσμπουργκ θα είναι σημαντική ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε ε, τι ε, δεσμεύσει ε, που αναλάβαμε τον Απρίλιο και πώς αυτές υλοποιούνται για τις πιο φτωχές χώρες. Θα φροντίσω να προετοιμαστεί στο ακέραιο αυτή η σύνοδος έτσι ώστε τα θέματα ανάπτυξης να κυριαρχήσουν στη σκέψη των ηγετών του G20. Δεύτερη σημαντική πρόκληση είναι η Επικείμενε διαπραγματεύσεις για να έχουμε το Δεκέμβριο στην Κοπεχάγη μια φιλόδοξη συμφωνία. Τα θέματα τα οικονομικά και του επιμερισμού του φόρτου είναι τα δύο σημαντικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουμε και εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε και πλήρω να ενταχθεί στη συζήτηση η ανάπτυξη. Στη συνέχεια, η πολιτική ανάπτυξη ίδια έχει προκλήσεις χωριστέ να αντιμετωπίσει. Εδώ μιλώ για τον όγκο τη βοήθεια, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια ή ακόμα και οι στόχοι τη χιλιετία για την ανάπτυξη, που είναι και αυτή η πρόκληση. Ε, το Νοέμβριο έχουμε μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χάσουμε στο λεγόμενο Κάγκρα, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, μπορέσει πριν το 2010 να έχει αποφασιστική σημασία. Το 2010 γνωρίζετε ότι είναι ένας ενδιάμεσος στόχος για ε, τις δεσμεύσεις του Γκλεν Ίγκελ της χιλιετίας. Είναι σαφές ότι θα πρέπει η Ένωση όχι απλώς να αυξήσει τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά ε, υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί αυτή ε, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ε, αν βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Ο κάτοχος μου συνήθιζε να λέει ότι δεν κάνετε απολεγγύη κάντε τουλάχιστον από συμφέρον. Και συμφωνώ απολύτως με την ανάλυση αυτή. Όταν σπανίζουν οι πόροι παντού, η ε, αποτελεσματική τους χρήση είναι εκ των ουκάνευ. Ο κώδικας συμπεριφοράς ε, για τον επιμερισμό εργασίας που πρόπερσε δέχτηκε το Συμβούλιο εφαρμόστηκε με τρόπο πάρα πολύ κατακαιρματισμένο, για να μην πω τίποτα χειρότερο μέχρι σήμερα. Ε, στόχος μου είναι να δώσω νέα όθηση στο θέμα αυτό τους επόμενους μήνες. Σε όλους τους τομείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαδραμάτισε πάντα ένα ρόλο ηγετικό και θα συνεχίσει να το πράττει. Βεβαίω, προσβλέπω στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη δική σα δηλαδή, για να πιέσουμε τα κράτη-μέλη. Στο ίδιο πνεύμα, ελπίζω να προωθήσω το θέμα τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση και η κλιματική αλλαγή ενισχύουν ακόμα περισσότερο αυτή τη βασική ανάγκη για περισσότερη συνέπεια. Στόχος μου είναι σύντομα να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτό το τομέα και επίση να ξεπεράσουμε τις δηλώσεις καλών προθέσεων. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να έχω σε βάθος συζήτηση με τους Ευρωπαίους Υπουργούς ε, Ανάπτυξης το Νοέμβριο. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, οι ίδιες οι χώρες ε, οι αναπτυσσόμενες θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά που τους αναλογεί, βελτιώνοντας τη διακυβέρνησή τους θα πρέπει ε, αυτό να γίνεται και με τρόπο διαφανή. Και εμεί ω δωρητέ έχουμε βασική ευθύνη να βοηθήσουμε του εταίρου μα να αναπτύξουν τη δυνατότητα διακυβέρνησή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την προσέγγιση αυτή με ε, διάλογο γενικό και τομεακό ενισχυμένο και με κίνητρα. Ένα πριμ αποτελεσματικότητα. ας πούμε. Στα τέλη του έτους θα αναθεωρήσουμε όλες τις στρατηγικές αναχώρα για να τις προσαρμόσουμε στη νέα κατάσταση. Αυτό ταυτόχρονα μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε τις δεσμεύσει και τις υλοποίησεις ε, στις χώρες και για να βελτιωθούν οι δομές της διακυβέρνησής τους. Από γεωγραφικής πλευράς τώρα θα εξακολουθώ να δίνω ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες και τις περιφέρειες που είναι πιο εύθραυστη κατάσταση, έχουμε δύσκολες εκλογές, όπως είναι η ε, ακτήρα Λεφαντοστού, η Γινέα Κόνακρη, ε, ο Νίγηρας, η περιοχή των μεγάλων ρυθμών, λιμνών, Μαδαγασκάρη, το κέρας της Αφρικής Ζιμπάμπουε, αλλά και ε, τα νησιά Φίντζη, ακόμα η Κούβα και αυτά είναι λίγα μόνα παραδείγματα. Στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό θέλω να έχουμε ενεργητική συμμετοχή για να σταματήσει ε, αυτή η κατάσταση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και το λαθρεμπόριο των ορυκτών πόρων που γίνεται και από δίκτυα μάλιστα ε, εγκληματικά. Ε, τέλος, η Υπουργική Τρόικα Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής τον Οκτώβριο θα είναι ευκαιρία να έχουμε μια ενδιάμεση αξιολόγηση των στόχων της Λισαβόνας του 2007. Αυτή η στρατηγική ε, είναι σε καλό δρόμο με συγκεκριμένα αποτελέσματα ήδη, αλλά θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο πολιτική όθηση έτσι ώστε ε, να διατηρήσουμε την πλήρη κινητοποίηση όλων των κρατών ευρωπαϊκών και αφρικανικών. Αυτό θα μας βοηθήσει να προετοιμάσουμε το έδαφος για ε, την επόμενη Σύνοδο Κορυφής Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, τέλος θα ήθελα να πω μερικά λόγια σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια που είναι εξίσου σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου μου. Και εδώ ε, έχω κληρονομήσει ένα μεγάλο πολιτικό πλαίσιο με Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια που εγκρίθηκε το 2007. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει εδώ ένα ρόλο κλειδί στην εκπόνηση αυτής της μεγάλης ε, διακήρυξης πολιτικής για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ελπίζω αυτή η καταπληκτική συνεργασία να μπορέσει να συνεχιστεί. Ορισμός νέου εισηγητού για ανθρωπιστικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τα άλλα θα βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα κλειδιά του επόμενου μήνε. Πρώτον, η διατήρηση του ανθρωπιστικού χώρου. Το 2008 122 ανθρωπιστικοί συνεργάτες ε, έχασαν τη ζωή τους σε όλο τον κόσμο. Μεγαλύτερος αριθμός από ποτέ. Δηλαδή είναι περισσότερο από ποτέ σημαντικό να φροντίσουμε η αποστολή τους να θεωρείται ως αμυγός ανθρωπιστική. Και αυτό θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από άλλες σκέψεις ε, γεωπολιτικές ή εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παραμένουμε ε, στη διάδοση και στη γνώση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Δεύτερον, ο προπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ανάγκε παραμένουν υψηλέ και όλο και περισσότερο αυξάνονται και με την κλιματική αλλαγή. Έχει τριπλασιαστεί ο ρυθμό των θεμενιών τα τελευταία δέκα χρόνια. Έτσι λοιπόν τους επόμενους μήνες με άλλους δωρητές θα συνεργαστούμε για να βρούμε μια συνολική λύση μεταξύ άλλων ε, με πρωτοβουλίες όπως το λεγόμενο Good Humanitarian Donorship και ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών. Τέλος, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή ε, μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων ανθρωπιστικών εργαλείων όπως είναι ας πούμε η πολιτική προστασία σε περίπτωση θεομηνίας. Έχει γίνει τεράστια πρόεδρος εδώ αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, μου δώσατε λίγο χρόνο και προσπάθησα να ε, ταυτοποιήσω τα πιο σημαντικά σημεία που θα χρειαστούν την προσοχή μου ως Επιτρόπου Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι οι ερωτήσει σας θα με βοηθήσουν σε συντομία ε, να μπω σε μεγαλύτερε λεπτομέρειε και να εξηγήσω. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω τη δέσμευσή μου ότι θέλω να προχωρήσω αυτά τα θέματα με ε, πίστη και αποφασιστικότητα. Όπω είπα στην αρχή τη παρέμβασή μου, το παρελθόν μου δείχνει ότι έχω και τα απαραίτητα προσόντα και την εμπειρία για να το πετύχω. Προσβλέπω σε αυτό στη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Mr. De Gift. Ευχαριστούμε κύριε Gift, λέει Πρόεδρος. Και τώρα θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Έχετε στη διάθεσή σας μισό λεπτό. Μισό λεπτό για μία ερώτηση προς τον υποψηφίο επίτροπο. Ε, θα υπάρξει υποβολή 4-5 ερωτήσεων και κατόπιν θα τις απαντήσει όλες όλες 4-5 ο υποψήφιος ε, επίτροπος και θα έχει 5 6 λεπτά στη διάθεση του για να απαντήσει. Πρώτος γύρος ερωτήσεων. Αλλά έχει δει σε διαδικαστικό. Κύριο Στάς. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Ναι, διαδικαστικό είναι. Είχε 15 λεπτά ο κύριος Φαν ε, ε, χρησιμοποίησε 12. Ελευθερώνονται 3 λεπτά. Απάντησε σε μερικές ερωτήσεις, αλλά και σε μερικές άλλες όχι. Την ερώτηση της κυρίας Τσίμερ από την ΚΟΕ, πολύ συγκεκριμένα. Αλλά και τη δική μου πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για τις προθέσεις τους. Ε, πόσο θέλει να μείνει, τρεις ε, μήνες, δώδεκα μήνες, μικρή περίοδο. ή θα ασκήσει πίεση για να το ανατεθεί το χαρτοφυλάκιο αυτό και στην επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Στασλή Πρόεδρε. Αυτό ήταν εναρκτήρια δήλωση, εισήγηση όπως ε, κάνουν όλοι και θα απαντήσει τις ερωτήσεις ε, ο υποψήφιος επίτροπος όποτε προβλέπεται. Δηλαδή μετά τον γύρο των ερωτήσεων. Συνεχίζουμε και δίνω τον λόγο στον κύριο Άλφ Βένσον του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική της ανάπτυξης ε, η διαφθορά. Διαπέστε μα ε, κύριε Τεχίου, τι συγκεκριμένα, τονίζω συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε να καταπολεμήσετε την διαφθορά, διότι γνωρίζουμε ότι είναι κάτι θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Δεύτερη ερώτηση τώρα να ακολουθήσει. Ενρική κύριε. S&D. Σοσιαλιστές. Bienvenido, señor Los efectos de la Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης αφορούν όλες τις χώρες του κόσμου και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως ε, ήταν ακόμα χειρότερη η κρίση για τις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις βιομηχανία Ανάπτυξη, ε, πίεση μεγάλη στους μετανάστες, πρώτες ύλε, εξωτερικό χρέος, με την ευκαιρία επομένως. Πολλές χώρες πέρασαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Έτσι έχουμε για τους φτωχούς ακόμα περισσότερη φτώχεια όμως. Τι λέτε κύριε Επίτροπε, δεσμεύεστε κάτι να κάνετε ώστε να κατανοήσετε αυτά τα προστατευτικά μέτρα τα οποία θεσπίζονται κατά των λιγότερων επιτυγμένων χωρών. I Πρόεδρος και τώρα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κέρνησε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω εγώ τι θα γίνει όσον αφορά την υπηρεαλιστική πολιτική της ε, Κίνας όσον αφορά την Αφρική. Εσείς θεωρείτε ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της στόχης και για την κονδυσιοναλιτέ. Δηλαδή τους όρους που επιβάλλει η Κίνα είναι επιβάλλει την μία αναγνώριση της Ταϊβάν. Θεωρείτε ότι παραβλάβουν τα μας από αυτή την πολιτική και αν ναι, τι προτείνετε να κάνετε. Κατρίν Κυρας, έχετε τον λόγο. Η χρηματοοικονομική κρίση παρόξενε τι ανισότητες. Αλλά οι ε, ανισότητες και στο ιστορικό της χώρας, αλλά και μεταξύ ημών και των χώρων μας ενδιαφέρουν. Οπότε έτσι δεν μπορούμε να ε, βοηθήσουμε την ανάπτυξη ούτε να προστατεύσουμε τους πιο φτωχούς από τα αποτέλεσματα αυτή τη ε, κρίση που εμεί ήδη δημιουργήσαμε. Εσεί από πλευρά Κομισιόν, τι μπορείτε να κάνετε για αυτή την κατάσταση, τι προτείνετε. Στα αγγλικά. Επίση, θα ήθελα να απαντήσετε πάνω σε αυτό που ρώτησε ο κύριο Στάση. Όσον αφορά το, το, την πτυχή του χαρτοφυλακίου σα που αφορά την ανάπτυξη. Πρώτα, σε ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο. Έχετε πέντε λεπτά. Eh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τέσσερις ερωτήσεις έγιναν. Μπορώ να πω ιστορίες ολόκληρες τώρα εγώ για αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις. Αρχίζω από τον κύριο Σπένσον για τη διαφθορά. Και ως υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου ασχολήθηκα με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, ποιος είναι ο βασικός λόγος της διαφθοράς και της ζωροδοκίας εκεί, γιατί δεν υπάρχουν πολλές πηγές εισοδήματος. Είναι και θέμα οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη νομίζω μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εκεί. Με ποιον τρόπο ε, πολύ στοχευμένα να δράμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Όταν ενισχύεται ο προπολογισμό των χωρών, πούμε, που είναι περίπου το μισό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη, η μακροοικονομική βοήθεια, να τη χρησιμοποιούμε για την προώθηση της καλής διακυβέρνησης των κρατών αυτών. Και να το συνδέουμε, ας πούμε, με όρους, με ε, χρηματικού ελέγχους. χρηματοπιστωτικού ελέγχου. Και έτσι έχει νόημα η μακροοικονομική βοήθεια από αυτή τη σκοπιά. Και κατά τα άλλα θα πρέπει να φροντίσουμε η δική μας αναπτυξιακή βοήθεια να μην ε, αφήνει να πάρει σφρή διαφθορά. Πάντως δεν υπάρχει εκεί πρόβλημα, είμαι αρκετά ήσυχο γι' αυτό. Το δεύτερο, κάτι που ρώτησε ο κύριος Γκερέρο για τον προστατευτισμό. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους τελικά δεν καταφέραμε ε, να ολοκληρώσουμε το γύρο της Ντόχα ήταν η αλληλεγγύη με τον τρίτο κόσμο. Όχι μόνο του πρώτου κόσμου με τον τρίτο, αλλά και μεταξύ των χωρών του Νότου, για να το πω έτσι, όπου δεν είχαμε πολύ μεγάλη σύμπνοια και συμπόνια για τις πιο φτωχές χώρες. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος προστατευτισμού που είναι μεγαδινό, αλλά από μόνο του ο προστατευτισμός δεν είναι η λύση. Θα πρέπει να δούμε και με τις αναπτυσσόμενες χώρες πώς θα τις βοηθήσουμε να χειραφετηθούν και να συμμετέχουν πλήρως στο διεθνέ εμπόριο. Aid for trade ας πούμε, βοήθεια για το εμπόριο. Είναι πάρα πολύ κεντρικό ζήτημα αυτό για μένα, να υπάρχουν και ε, ποιοτικά προϊόντα εξαγωγών από τις χώρες αυτές γιατί από μόνος του ο προστατευτισμός δεν απαντά. Απαντώ στο Σαλ Γκέρν στα γαλλικά για την Κίνα. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και περίπλοκο ταυτόχρονα. Διότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε ε, αμυγός και μονομερός αρνητικοί. Η Κίνα μπορεί να φέρει πολύ σημαντικά κονδύλια στην ανάπτυξη της Αφρικής, για παράδειγμα, αλλά εκεί χρειάζεται ένα αυστηρό διεθνές πλαίσιο και επίσης να σέβεται η αυτό το διεθνές πλαίσιο. Και εκεί πραγματικά το πρόβλημα είναι ακαθόδες. Βράχει πρόθεσμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ με τις κινέζικες επεμβάσεις είναι η δική μας κυρίως αντίδραση. Τι διαπίστωσα επανειλημμένα. Ακριβώς επειδή η Κίνα το σε κάποια χώρα, ξαφνικά η στάση ορισμένων κρατών μελών απέναντι στη χώρα αυτή άλλαζε. Και είχαμε την εντύπωση ότι επανέρχεται ο ψυχρός πόλεμος. Ότι σε ορισμένες αφρικανικές χώρες ήταν όλα δυνατά. Γιατί θεωρούσαμε ότι έχει στρατηγικό συμφέρον κάποιος. Λοιπόν, μην κοιτάμε μόνο την Κίνα, να κοιτάμε και τι κάνουμε και εμεί οι ίδιοι κυρίως. Να κοιτάμε και στον καθρέφτη καμιά φορά. Κυρία Γκρέζ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω την ερώτηση του κυρίου Στά. κανένα. Εμένα με όρισαν ως ε, Επίτροπο Ανάπτυξης τώρα, φαντάζομαι ότι ο κύριος Στάς θα είχε δυσκολίες να πει ότι τα πέντε χρόνια ω υπουργό Εξωτερικών δεν ασχολήθηκα με τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Και βέβαια ενδιαφέρομαι ειλικρινά για το φάκελο αυτό. Θα εξερθεί από την κατανομή των χαρτοφυλακίων στην επόμενη επιτροπή, σε εφόσον επιβιώσω σήμερα. Thank you. We will now start... Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερώτα απαντήσεων. Το λόγο έχει η συνεργαζόμενη επιτροπή, ο αντιπρόεδρος της, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Φιωρέλο. Έκανα λάθος. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, είμαστε στο δεύτερο γύρο. Διάστηκα υπερβολικά. Ο κύριος Ντέβα έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νόμιζα ότι με παρασύρατε με τη διασύνη αυτή. Θέλουμε να ρωτήσουμε τον Επίτροπο. Έχετε πολύ σοβαρό έργο στα χέρια σας. Εφόσον πρέπει να φέρετε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες. Στην ανάπτυξη, ο τομέας αυτός είναι από τους πιο απλούς όπου μπορούμε πραγματικά το έργο μας να το πάμε κοντά στους πολίτες. Διότι οι πολίτε μπορεί να εγκρίνουν αυτά που κάνουμε και να μην υπάρχει και καμία διαφωνία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο τη συνθήκη τη Λισαβόνα. διότι με το δημοψήφισμα για τη συνθήκη τη Λισαβόνα, συζητήσαμε πολύ το κατά πόσον πρέπει η Λισαβόνα να πάει πολύ πιο κοντά στο δικό μα το έργο και να προσεγγιστεί. Το 2002 όμω, είπατε στην Πλάμπρα ότι η συνταγματική συνθήκη θα πρέπει να είναι πιο εύληπτη και ότι ο στόχος της συνθήκης της Λισαβόνας φαίνεται να είναι δυσανάγνωστη. Θεσμικά λοιπόν, ενώ οι συνθήκε κανονικά έπρεπε να είναι σαφεί, αυτή η συνθήκη στόχο είναι να είναι ασαφή. Αυτή είναι η επιτυχία τη. Εδώ βλέπω μια αντίφαση με την ε, πρόθεσή μας να φέρουμε τα πράγματα πιο κοντά στου ανθρώπου, στου πολίτε. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Σίμερ. Την περασμένη θητεία ως Επιτροπή αλλά και ως πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχοληθήκαμε επανειλημμένα με τους στόχους χιλιετίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους. Ξέρουμε ότι απέχουμε πόρο από την υλοποίηση. Εμένα με ενδιαφέρει σημαντικό και συγκεκριμένο εργαλείο που έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τώρα θεωρούμε ότι έχει ε, χρησιμοποιηθεί με τρόπο πάρα πολύ ανεπαρκή. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τι κάνετε εκεί. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε να δοθεί εντολή από τις χώρες μέλη για να είναι αποτελεσματική η αναπτυξιακή βοήθεια και οι πιστώσεις πραγματικά στοχευμένες. Thank Ευχαριστούμε. Και τώρα η ομάδα της Ευρώπης της ε, Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Παρακαλώ. Όχι. Τότε ο κύριος Φρανκ Φανέκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντεχιούχτ, ένας Ευρωπαίος Επίτροπος θα πρέπει να είναι περάνω πάση υποψίας ε, διαπλοκή συμφερόντων και διαφθοράς. Εσείς ε, δεν είστε υπεράνω. Ε, σας έχουν πιάσει στα πράσα με την κρίση της φόρτης. Είχατε την παραμονή της κατάρρευσης της τράπεζας επαφή και τηλεφωνική, εσείς με το διευθυντή της τραπέζης, αυτό έχει αποδειχθεί. Το ξέχασε ο Υπουργός. Την παραμονή συζήτησε, ε, τηλεφωνήθηκε και τα μέλη της οικογένειας του πουλούσαν τεράστιες ε, ποσότητες μετοχών στην αγορά. Όλα αυτά είναι τελείως αναξιόπιστα. Φοβάμαι ότι δεν προσφέρεστε για να λάβετε πόστο αυτό ε, του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Είστε τελείως ακατάλληλος άνθρωπος σε τέτοια θέματα που είναι τόσο ευαίσθητα για τη διαφθορά. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Um, Mr. Mr. Deva, um, I think I know... Κύριε νομίζω ότι ξέρω για ποια δήλωση και συνέντευξη μιλάτε. Αν και δεν την έχω μπροστά μου. Έχω μια ολόκληρη συλλογή, αλλά όχι αυτό. Αυτό που εννοούσα νομίζω και αληθεύει είναι ότι με τη σταγματική συνθήκη προσπαθήσαμε να έχουμε ένα πολύ κατανοητό κείμενο συνθήκης. Ξεκινώντας από την εικασία ότι αν είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει κανεί και θα το διαβάσουν οι πολίτες και θα το καταλάβουν. Αυτό που συνέβη είναι ότι σε καμία περίπτωση τη διάβασαν και δεν κατάλαβαν το παραμικρό. Επίσης αληθεύει ότι όταν έγιναν συζητήσεις για το πώς θα διορθώσουμε τις αποτυχίες που είχαμε με τη συνταγματική συνθήκη στη Γαλλία και την Ολλανδία, υπήρξε μία μετατόπιση εγώ υπήρξα μάρτυρα τη μετατόπιση και μέρο τη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μια μετατόπιση να περάσουμε σε κάτι που να είναι τεχνικό τουλάχιστον ορθό και η συνθήκη τη Λισαβόνα είναι, αλλά ιδιαίτερα περίπλοκο. Κατά τρόπο ώστε να μην να μπορεί να γίνει συζήτηση για αυτό το κείμενο. Αυτό ήταν η θελημένη ε, απόφαση του και πρόθεση του Συμβουλίου. Όσο και αν επικρίθηκε, είναι γεγονό. Συνέβη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήταν η απόκριση στι αποτυχίε τη πολιτική διαφάνεια ανοιχτών ε, πυλών που είχαμε εφαρμόσει με τη συνταγματική συνθήκη. Να λοιπόν η απάντηση για τα προβλήματα που μπορούμε να δούμε σε μερικέ εβδομάδε. Κύριε Βανέκε, θα με εξέπλητε να με θεωρούσατε ικανό για τη θέση αυτή και ότι θα μου άρμοζε. Και αν το λέτε εσείς, ε, ε, δηλαδή αν με θεωρούσετε κατάλληλο κάτι θα πήγαινε πολύ στραβά, είτε με εσάς είτε με μένα. Το ότι με θεωρείτε απολύτως ακατάλληλο ε, το θεωρώ φυσιολογικό και ούτε με ανησυχεί καθόλου. Αλλά ε, θα με εξέπλητε επίσης που κάνετε ερώτηση, παρατήρηση και όταν τα κάνετε αυτά να σέβεστε και την αλήθεια, έτσι. Και αυτό θα ήταν τελείως ε, πρωτοτυπία σε ό,τι σας αφορά. Εγώ δεν σας διάκοψα κατά τα άλλα. Αν κοιτάξετε το φάκελο, που μπορεί να μην το κοιτάξατε ή και να το κοιτάξατε, θα διαπιστώσετε ότι γράφει επιλέξει ότι μίλησα με το διευθυντή ε, του υποκαταστήματος τον Μπελάρε, όχι στις Βρυξέλλες, και μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει καμία πώληση μετοχών. Και έχει γίνει έρευνα ε, στο θέμα αυτό από το εφετείο της Γάνδης που λέει και με επενεί πολύ ε, στο Βελίο γιατί ο κύριος Χέιμανς ακριβώς ξεκίνησε και την έρευνα και την ανάκρισή μου και έχει ε, ασχοληθεί με όλο το φάκελο του θέματος φόρτης και δεν μπορεί να μου προσάψει κανείς το παραμικρό, ούτε υποψία, ούτε τίποτα διαφορετικό. Στα γαλλικά τώρα. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ιδιαίτερος σε αυτέ τις προσπάθειες, διότι ασχολείται με τη διευκόλυνση των χρηματοδοτήσεων των ε, χωρών ΑΚΕΠ. Επίσης, το Ταμείο για, την, ε, για τη Διάρθρωση δημιουργήθηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που καταφέρνει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη. Για κάθε ευρώ που κερδίζουμε από τις ε, επενδύσεις αυτές τα, διαθέτουμε στην ανάπτυξη για τις υποδομές. Υποδομές ε, οικονομικές, γεωνομικές, εξυγίανση υδάτων και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως ένα γενικό πρόβλημα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό είναι ότι υπάρχει και ένα όριο στις, στους πόρους της. Ε, οι πόροι είναι περιορισμένοι για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα έπρεπε να αυξήσουν το αποθεματικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά τρόπο ώστε να μπορεί να διαθέσει περισσότερα και μάλιστα κατά τρόπο κατεπήγοντα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει λύση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως προς τον τρόπο λειτουργία της και τη δομή της λύση που να αλλάξει κάπως τα πράγματα να γίνει δηλαδή λίγο διαφορετικά, διαφορετική λειτουργία της από τους θεσμούς του Bretton Woods. Γιατί τώρα λειτουργεί κατά αυτό το πρότυπο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε λοιπόν να κάνει πολύ περισσότερα και είναι και αναγκαίο όπως πολύ σωστά έχετε παρατηρήσει. <coughs> Ευχαριστούμε κύριε Τεγκούχτ. Τώρα θα δώσω το λόγο στις ε, συναρμόδιες επιτροπές πρώτα πρώτα ο πρόεδρος της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων για 45 δευτερόλεπτα κύριο Πιοβέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Δευτέρου 2009 ενέκρινε ένα ψήφισμα όσον αφορά την Γάζα και την ανθρωπιστική κατάσταση. Εκεί ζητούσε το Κοινοβούλιο, στο τρίτο σημείο, να προχωρήσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο υπολογισμό των ε, ζημιών που υπάρχουν εκεί και επίσης ε, να υπάρξει μια αξιολόγηση γενικότερη εις βάθος των αναγκών του, του, του πληθυσμού, τόσο ώστε να προχωρήσουμε σε ανασυγκρότηση πέρα τη ε, παράθεση και λαμβανόμενο όψη ότι εμείς είμαστε ο βασικός δανειστής και δωρητή ε, πάνω από 135 εκατομμύρια έχοντας το 2008, 430 συγγνώμη, και είχαμε άλλα 80 εκατομμύρια που προβλέπονται ήδη για το 2009 και αυτά τα 439 εκατομμύρια τα οποία αποφασίστηκε να δοθούν στο, στη διεθνή ε, διάσκεψη της Δευτέρας Τρίτου του 2009 ε, νομίζω ότι θέλει όλος ο κόσμος να μάθει ακριβώς πού καταλήγει αυτή η υπόθεση της ε, αξιολόγησης. να μας προτίθεστε στους εμείς επόμενους μήνες να συνομιλήσετε μαζί μας. Το κόβει το, το, το μικρόφωνο η πρόεδρος διότι έγινε υπέρβαση του χρόνου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, που είναι η κυρία Χάιντι Χάουταλα, η οποία είναι η πρόεδρο τη Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχετε το λόγο για 45 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ να κινηθείτε στα χρονικά πλαίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, κυρία Χάουταλα. Βεβαίω και θα το πράξω αυτό. Εμεί έχουμε πάρα πολλέ υποχρεώσει όσον αφορά τη, τη, την Ευρωπαϊκή Συνένεση για το mainstreaming τη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ερώτηση μου είναι η εξή, κύριε υποψήφιο. Πώ θα εξασφαλίσετε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θα πρετανεύσουν στην προσέγγισή σας για την πολιτική που θα ασκήσετε και πώς θα εξασφαλίσετε ότι και στη φάση της εκτέλεξης ακριβώς όσον αφορά και την ισονομική στήριξη θα ισχύσει το ίδιο. Διότι νομίζω ότι αυτό το mainstream των δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ βασικό για πάσα δράση εξωτερικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και δίνει το λόγο τώρα στον κύριο Ντεχίχ. Έχετε το λόγο για 3,5 με τέσσερα λεπτά. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, νομίζω ότι όντως είναι μια τεράστια ανθρωπιστική πρόκληση. Αναφέρεστε σε μια έρευνα που αποκάλυψε πολλά πράγματα. Η κατάσταση στη Γάζα ε, μου είναι γνωστή και στη Δυτική Όχθη κατά τα άλλα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που προβληματίζει τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ. Διότι το Ισραήλ ουσιαστικά δεν συνεργάζεται για την ανθρωπιστική βοήθεια και προσπαθεί μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας να ε, αντιδρά και τη, περιορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Επανειλημμένα έχουμε πει να ανοίξουν μεθοριακή σταθμή με τη Γάζα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα προϊόντα να μπορούν να εισάγονται. Ο κατάλογος των προϊόντων να διαφρυνθεί. Τώρα είναι πάρα πολύ λίγα, πάρα πολύ περιοριστικά. Και για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν αφήνουν να περάσουν τα προϊόντα στη Γάζα και δεν μιλώ για άλλα ε, σημαντικά, για το τσιμέντο, ας πούμε, για την ανασυγκρότηση. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μήνες ολόκληρους μετά την καταστροφή δεν μπορούμε να βάλουμε τσιμέντο στη Γάζα. Για να χτίσουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους ξανά. Νομίζω ότι η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί και ακόμα περισσότερα. Και εκεί είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις και Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί ε, με κυβερνητικέ οργανώσει, τα Ηνωμένα Έθνη, αναπτυξιακοί εταίροι με του οποίου συνεργαζόμαστε σε επτά τομεί. Ε, ε, διατροφή, στέγαση, ίδρυυση, κοινωνική υποστήριξη, προστασία και συντονισμός. Κάθε χρόνο αυξάνεται η χρηματοδότηση. Κατά τα άλλα, και ο αρμόδιος επίτροπος για την ανάπτυξη αλλά και για τις εξωτερικές σχέσεις συνεργάζονται ε, και με τρόπο εφάνταστο βρίσκουν και νέα κονδύλια. Και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η Γάζα επιβιώνει λόγω της ευρωπαϊκής υποστήριξης, χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη. Είναι γεγονός αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, καταρχάς πιστεύω ότι το σημαντικότερο δικαίωμα στα αναπτυσσόμενα κράτη είναι να εκριζωθεί η απόλυτη ένδυα. Αυτό είναι το υπαριθμό ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή να μπορεί ο κόσμος να τρέφεται με τρόπο αξιοπρεπή. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι σε πολλές ε, περιοχές ε, καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε από τις χώρες, είτε από πολιτοφυλακές. Στο Ανατολικό Κονγκό, για παράδειγμα, ο Μισελ και εγώ το γνωρίζουμε πολύ καλά, υπάρχουν τεράστιες βιαιότητες, ε, σεξουαλικά εγκλήματα. Είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι μόνο παραβίαση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι άρνηση κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί καλή στα κανείς με τη μακροοικονομική βοήθεια να κάνει θετικά βήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και υποστηρίζοντας συγκεκριμένα έργα, projects. Η μακροοικονομική βοήθεια θα πρέπει να προσαρμόζεται πολύ συγκεκριμένα ε, και αυτό μας βοηθάει να έχουμε περισσότερα μέσα για να γίνονται ε, ε, πολύ ενεργή και πολύ εντατική πολιτική διάλογη. Αλλά όταν υπάρχουν και προβλήματα θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα της μακροοικονομικής βοήθειας. Με τη Ρουάντα, ας πούμε, είχαμε ε, πρόβλημα, όπου η Ολλανδία και η Σουηδία, αν δεν απατώμε, και το ε, Ηνωμένο Βασίλειο μεσολάβησαν και αναδιπλώθηκε η Ρουάντα και τα μάζεψε. Θα σα δώσω και στη συνέχεια το λόγο να συνεχίσετε, λέει η πρόεδρο που διακόπτει τον κύριο Ντεχόχτ. Αρχίζει τώρα ο τέταρτο γύρο ερωτήσεων ε, των μελών. Ο κύριο Γκέι Μίτσελ, παρακαλώ. you, uh, I... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα από την ενοποιημένη εκδοχή τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία τη, στην οποία την οποία παραθέσαμε προηγουμένως για την αναπτυξιακή βοήθεια, λέει στο άρθρο 2 8.2 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα σέβονται τι δεσμεύσει και θα λαμβάνουν υπόψη του στόχου που εγκρίθηκαν στο επίπεδο του ΟΗΕ και άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών. Στο άρθρο 211 μιλάμε για τη συμπληρωματικότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της ένωσης και των κρατών μελών που θα συντονίζουν τις πολιτικές τους για την αναπτυξιακή βοήθεια μετά από διαβουλεύσεις. Τι βήματα λοιπόν θα λάβετε εσείς για να είσαστε βέβαιοι ότι τα δύο αυτά εδάφια θα γίνουν σεβαστά. Και ιδιαίτερος Πώ θα ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να νομοθετήσουν ε, πάντοτε ε, ε, με ένα δραστικό τρόπο για να καταφέρουν το ποσοστό του 0,07%. Κάποια κράτη-μέλη υπερβαίνουν τη δέσμευση αυτή, κάποιοι άλλοι δεν την λαμβάνουν καν υπόψη και χρησιμοποιούν το απόθεμα αυτό για χώρια χρήση. Τι θα κάνετε αυτό και πώ θα διασφαλίσετε εδώ το συντονισμό. κύριος Ντάβιντ Μαρία Σασόλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχει υποτιμηθεί το πρόβλημα Τη Ανατολή, και θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε και τη δέσκεψη των κλιματικών αλλαγών στην Κοπενχάγη. Σκεφτείτε το θέμα τη μείωση των εκπομπών που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καταπολέμηση της ε, αποψήλωση των δασών. Ε, είναι ένα ζήτημα σημαντικό και αυτό και σκεφτείτε ότι αυτό είναι πάντοτε μια δίκαια που διαπράττουν τα πλούσια κράτη ει βάρο των αναπτυσσόμενων χωρών. Επίση, θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσει, επενδύσει στην τεχνολογία, στη μείωση των εκπομπών ε, του διοξιδίου του άνθρακα, επίσης την αιωλική ενέργεια, την κατακράτηση άνθρακα. Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή σχετικά και ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια ήταν ε, πολύ σωστό που και εσείς το θυμήσατε ως προτεραιότητά μας επειδή με Ιταλός θα ξέρετε ότι μας είναι προσφυλές, αυτό είναι σημαντικό τι γίνεται με την εκδίωξη των λαθρομεταναστών και των παράνομων με συγχωρείτε σας διακόπτω το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι εξίσω εύστοχο, αλλά και ίσω και περιττό. Αφορά την συνοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντεκούρτ ε, τι σκοπεύει να κάνει σε περίπτωση που στο επίπεδο της Επιτροπής άλλη επιτροπή, επιτροπή θα τον εμποδίσουν να ακολουθήσει μια συστηματική προσέγγιση θα ήθελα να μας δείτε στη διάσκεψή μας όταν θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και άλλες παζοκεφαλιές στους ε, άλλους επιτρόπους και τι θα κάνετε εσείς αν εκείνοι προσπαθήσουν να σας βάλουμε τη σειρά τους τρικλοποδιά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει τη Κοπενχάγη, πώ σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι και οι στόχοι περί κλίματος ε, θα επιτευχθούν, όπω και τα δικαιώματα στην ανάπτυξη θα διασφαλιστούν για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και πώ θα βεβαιωθείτε ότι το Ταμείο για την προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ θα συνδυαστεί με τι ανάγκε τη αναπτυξιακή βοήθεια, ODA. Επίτροπε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Eh, ναι, κύριε Μίτσελ. Ο στόχος του 0,7% είναι βέβαια πρόκληση για κάθε κράτος μέλος. Εγώ προέρχομαι από ένα κράτος μέλος που πιστεύω σέβεται αυτό το στόχο, αλλά σε κάθε ζήτηση για τον προπολογισμό βλέπω να επανέρχεται αυτό το θέμα επιτάπιος το και συζήτηση. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίοδους οικονομικής κρίσης να μην μειώνονται αυτομάτως ε, τα ποσά αλλά και τα ποσοστά για το ΑΕΠ. Θα πρέπει ας πούμε, να βρίσκουμε τρόπους και τεχνητούς να φτάνουμε στο 0,7 όπως είναι η διαγραφή του χρέους. Ας πούμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το φροντίσει πολύ αυτό και αν χρειάζεται να κατονομάζει και να στιγματίζει και να ε, διαπομπεύει name and shame τις χώρες αυτές. Και μπορεί να δώσει και συμβουλές και εντολές στα κράτη-μέλη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ε, έτσι, και πρωτοπόρο. Έγιναν δύο ερωτήσεις για την Κοπεχάγη τώρα. Δύο είναι τα σημαντικά θέματα ε, στην Κοπενχάγη. Ε, οι δεσμεύσει μα για τις εκπομπές, αλλά τουλάχιστον εξίσου σημαντικό είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Όχι μόνο στον αναπτυγμένο κόσμο, αλλά και ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και είναι προφανέ ότι ο αναπτυγμένος κόσμος θα πρέπει να βοηθήσει και τον αναπτυσσόμενο με τη χρηματοδότηση. Εκεί πραγματικά μιλάμε για τεράστια ποσά. 250-500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι οι υπολογισμοί. Ακόμα και αν πάρει το χαμηλότερο το 250 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, διαρωτώ με πώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Το χρόνο, έτσι. Από το εμπόριο ε, των εκπομπών, ε, των δικαιωμάτων, εντάξει, το μεγαλύτερο ποσοστό. Έχω την εντύπωση όμως, βεβαίω μπορεί και να σφάλω, ότι ο αναπτυσμένο κόσμο θεωρεί ότι μπορεί να ε, ξεπληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τις αγοραπολισίες των εκπομπών, χωρίς να μειώνει τις ε, εκπομπές. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε αυτά τα τεράστια ποσά ε, να δαπανώνται σωστά και να αξιοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν δούμε τι τεράστια προβλήματα υπάρχουν από τώρα με τα διαθέσιμα ποσά, μπορούμε να μιλάμε για 80 δισεκατομμύρια το χρόνο. Επί τρία, για αυτό που σας έλεγα. Υπάρχει και κάποια θέμα εκεί αποφροφητικότητας από τα αναπτυσσόμενα κράτη και μεγάλο. Σάρλα Γκέρενς, σε ευγνωμονώ που θα με βοηθήσεις. Ε, και να μου βάλεις παζοκεφαλιές και εμένα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να με στριμώχνεις. Ελπίζω να μην το κάνεις όμως. Και ε, ελπίζω ότι ε, όλη η Επιτροπή Ελπίζω μάλλον να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η αναπτυξιακή συνεργασία και η πολιτική είναι σημαντική για την επιβίωση την ίδια της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη ελεγγύη και στην Επιτροπή σας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. We will now start the fifth round. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε τον πέμπτο γύρο ερωταπαντήσεων τώρα για τα μέλη της Επιτροπής μας πάλι. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει ένα ρητό που λέει, μη δίνετε ψάρια σε αυτόν που πεινάει, δώστε του ένα καλάμι για ψάρεμα. Τι εννοούμε λοιπόν με την ελάφρυνση της ένδυας. Μπορεί να εννοούμε και δημιουργία πλούτου τελικά κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα λοιπόν μια πιο συγκεκριμένη απάντηση γι' αυτό. Τι προγράμματα δημιουργίας πλούτου, παραγωγής πλούτου έχετε υπόψη σας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. The floor is for Madame Michel. Το ρόλο έχει η κυρία Στίφλερ. Oui, donc le consensus... Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Αναπτυξιακή Βοήθεια συνυπεγράφει από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2007. Τι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε λοιπόν για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Τι θα κάνετε κατά τη θητεία σας για να φέρετε εις πέρα στι δεσμεύσει που αναλήφθησαν για τη δράση αυτή, ιδίω για την κινητοποίηση περαιτέρω χρηματοδότηση για τι αυξανόμενε ανθρωπιστικέ ανάγκε. Το λόγο ο κύριος έχει ο κύριος Νόισερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντεχέχτ, είπατε και σημείωσα ότι είστε πρόθυμος να συνεχίσετε την πολιτική κληρονομιά που αναλάβετε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ερωτώ, τι γίνεται με τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις διακοιμάσεις των τιμών των τροφίμων και τις επιπτώσεις ε, της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε πολλές φτωχές χώρες. Ποιες δυνατότητες πιστεύετε έχει και ποιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κινητοποίηση και ε, νέων κονδυλίων για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ευχαριστώ. Πάλι ο κύριος Γκέρενς. Όχι, όχι. C'est pas. D'accord. Alors, donc, il y a un changement. D'accord. C'est pour M. Ivo Ο κύριο Ιβο Βάγκελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω το εξή ερώτημα. Τι δυνατότητες ε, θεωρείτε ότι υπάρχουν τόσο ώστε να μπορέσουμε ε, όσον αφορά τη συνεργασία με την Αφρική, να προωθήσουμε την περιφερειακή συνεργασία. Επίσης, για τον Ταρφούρ, τι προτίθεστε να κάνετε. Merci. La parole est... Ευχαριστούμε. Το λόγο θα κυρίως Γέρενς τελικά. Non, parce que c'est encore là. Ο κύριο Βάγκερ έλαβε το λόγο στη θέση του κύριου Μα πάλι Γκέρεν γράφει εδώ. So uh, και αυτό το δεύτερο γύρο. Ο επίτροπο έχει το λόγο για να απαντήσει σε πέντε λεπτά. Mr. Um, Diva, I think you... Κύριε Δίβα, αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό για την παραγωγή πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εδώ πρέπει να αναλάβουν σημαντικό ρόλο. Και το ιδιωτικό επιχειρήν δεν είναι μόνο οι άμεσες επενδύσεις, δεν εννοώ μόνο αυτό. Δεν εννοώ μόνο ευρωπαϊκέ και αμερικανικέ εταιρείε που θα αναλάβουν δράση στι αναπτυσσόμενε χώρε. Εννοώ πώ να αναπτύξουμε, να προωθήσουμε τη μεσαία τάξη σε αυτές τις χώρες. Ιστορικώ, αυτό έχει συμβεί και σε άλλε περιοχέ του κόσμου και ξέρουμε ότι ο ρόλο τη τάξη αυτή είναι σημαντικό. Αν δημιουργηθούν συνθήκε που θα ευνοήσουν τη μεσαία τάξη, μέτρα όπω μακροπιστώσει, μεγάλε πιστώσει που είναι εδώ σημαντικέ, μικροπιστώσει επίση, δανεισμό χρήματος εμπορική βοήθεια, διότι και οι υποδομές στις χώρες αυτές είναι σημαντικές, πρόσβαση στις αγορές, διότι αν δεν έχει κανείς πρόσβαση δεν μπορεί να πάει στην αγορά. Ε, το πρόβλημα κάποιες φορές είναι ακόμη και σωματικό, υπαρκτό. Δεν υπάρχει απαραίτητη παραγωγικότητα. Και ο ρόλος των γυναικών εδώ, είναι σημαντικό. σημαντικός, διότι μένουν εκτό της οικονομίας ε, στι αναπτυσσόμενες χώρε οι γυναίκε και θα πρέπει να περάσει και στα χέρια του ένα μερίδιο τη αγοράς. Κυρία Στίφλερ, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη ανθρωπιστικής βοήθεια, αλήθεια είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερο αιτήσεις, περισσότερες αιτήσει για, για ανθρωπιστική βοήθεια και ανθρωπιστικές κρίσεις, ανθρωπογενείς ή από φυσικά αίτια. Διαπιστώνουμε ότι τα κονδύλια δεν αρκούν. Ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το σημαντικότερο παγκοσμίω προπολογισμό, κάπου 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίω, για του σκοπού αυτού. Θα πρέπει να δούμε σε, ποιο, σε τι βαθμό θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και τις διαδικασίες και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δωρητών. Όποτε υπάρχει ανθρωπιστική κρίση βλέπουμε ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας ε, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Και σε πρώτη φάση θα πρέπει να κοιτάξουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για τις κλιματικές αλλαγές, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς έδεσε το ερώτημα, δεν τον είδα γιατί είναι τόσο γοργός ο ρυθμός που δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις αλλαγές στην αίθουσα. Για τις κλιματικές λοιπόν αλλαγές, Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της χρηματοδότησης. Υπάρχει όμως και το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές του κόσμου αναπτυσσόμενες είναι σοβαρές οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, όπως στα νησιά. Τα ερχόμενα χρόνια λοιπόν θα έχουμε μάλλον μεγάλη ε, μεταναστευτικά κύματα λόγω των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό θα είναι ένα επιπλέον άχθος και για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις δικές μας βεβαίως. Μιλάμε για 300 εκατομμύρια ανθρώπων που μπορεί να πληγούν από τα κλιματικά φαινόμενα την ερχόμενη δεκαετία. Κύριε Δέγκλιο. Η περιφερειακή διάσταση είναι η διάσταση του μέλλοντος, ξέρετε. Θα πρέπει όμως να τολμούμε να πούμε ότι η περιφερειακή συνεργασία δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Αν δούμε κανείς στην, ε, στην Αφρική τι επικαλύψεις υπάρχουν σε μεγάλο περιφερειακές συνεργασίες. συνεργασίας, είναι πολλά κράτη-μέλη σε διαφορετικούς περιφερειακούς οργανισμούς και σε πιο αναπτυγμένα μέρη και στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Η περιφερειακή συνεργασία δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Το αντίθετο μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Συνεργασία επενδύει πολύ από το σημερινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Αν δεν απατώμε, προβλέπονται 2,8 δισεκατομμύρια για περιφερειακά έργα. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακριβώ μέχρι να επιτύχουμε αποτελέσματα. Η περιφερειακή συνεργασία έχει και ένα δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή, οι στοδιοινικές είναι ενδεχομένω ε, μία λύση ε, για να αποφεύγουμε πολιτικά προβλήματα μεταξύ κρατών. Ε, πολλά από τα σύνορα στην Αφρική είναι ευθείε γραμμές που έχουν χαρακτή και δεν είναι φυσικά σύνορα. Και αν υπάρχει περίπτωση να λυθούν από την περιφερειακή συνεργασία, πραγματικά ε, προλαμβάνει και κρίση σε αυτό. Και τώρα να αρχίσουμε τον έκτο γύρο ερωταπαντήσεων. Θα υποβάλει ερωτήσει η Συνομόδια Επιτροπή του Διεθνού Εμπορίου, κύριε Αρήφ από τη συντονιστή και τον λόγο. Σαν δευτερόλεπτα, κύριε Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα βιώνει ότι δύο δι ευρώ πρόκειται να διατεθούν για ε, βοήθεια στο, στον του εμπορίου. Όμω δεν μα λέει από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα. Θα είναι επιπλέον χρήματα, όπω έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επίση, το Κοινοβούλιο δεν έχει κανέναν έλεγχο όσον αφορά αυτά τα θέματα. Όλα αυτά δεν έχουν μπει στον προπολογισμό. Άρα, εμεί είμαστε πάρα πολύ ε, προβληματισμένοι για πώ θα γίνει αυτό. Γιατί αυτό αφορά και την ε, Επιτροπή Ανάπτυξη αλλά και το εμπόριο. Παρακαλώ, διασκεδάστε τι εμβολίε μα και πέστε μα ακριβώ πώ θα συνεργαστούν με του βουλευτέ οι υπηρεσίε για να μα δώσουν ό,τι πληροφορία χρειαζόμαστε και να μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ έχετε το λόγο για 45 δευτερόλεπτα. Κύριε Επίτροπε, αυτό το κύριο συζητάμε το προπολογισμό. Εσείς ε, έχετε ένα χαρτοφυλάκιο περιορισμένου χρόνου. Τι θα κάνετε με τα χρήματα για το Aid for Trade. Να είναι νέο χρήμα και όχι αναδιανομή παλαιών πόρων και είστε πρόθυμος να δώσετε συγκεκριμένες ημερομηνίε στο Κοινοβούλιο για ενημέρωση για το πώς ε, δαπανώνται αυτά τα κονδύλια ε, της βοήθειας για το εμπόριο, Aid for Trade. The floor is for the Commissioner designate to answer. Ο υποψήφιος επίτροπος έχει το λόγο για να απαντήσει στις δύο αυτές ερωτήσεις. Um, Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Πράγματι με τον προπολογισμό. και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης βεβαίως, διότι αυτό είναι, ένα, είναι μέρος των ε, κονδυλίων που μπορεί να δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν περνούν από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Εάν δει κανεί με προσοχή γιατί συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να δει τις κλίδες κατανομής πάνω απ' όλα λοιπόν το κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει πρώτο από όλου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Θα πρέπει και αυτό να περάσει στον συνολικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήμουν υπέρ αυτή τη αλλαγή. Το ερώτημα για την αναπτυξιακή βοήθεια Aid for Trade. Είναι σοβαρό το ποσό που διατίθεται στην περίπτωση του Aid for Trade στήριξη του εμπορίου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικότερο και από άλλες περιπτώσεις. Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με την ύπαρξη χρήματο, αλλά με οικονομικές ροές. Δεν ξέρω κατά πόσον εγώ θέμουν σε θέση εδώ να επηρεάσω την κατάσταση. Σημαντικό είναι ότι τα ποσά διαθέσιμα. Και αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι να έχουμε αρκετά προγράμματα και καλά προγράμματα ώστε να μπορούν να εκταμιευθούν τα κονδύλια αυτά. Το να δημιουργήσουμε έναν επιπλέον χρηματοδοτικό μηχανισμό για το Aid for Trade δεν μου φαίνεται πολύ ρεαλιστικό ως κίνηση. Θα πρέπει να ζήσουμε με το γεγονός ότι αυτό αποτελεί μέρος του, του FED, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και ότι ακριβώς αποτελεί μέρος των όσων προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τώρα τον 7ο γύρο ερωτήσεων για τα μέλη της Επιτροπής μας. Το λόγο έχει η κυρία Σαργαντίνη για τους πράσινους. Ξεκινήσατε με ένα απαράθεση από τον προκάτοχό σας. Αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη και δεν δράτε λόγω αλληλεγγύης, δράστε για το συμφέρον σας. Τι θα γίνει όμω με τι χώρε ΑΚΕ που έγραψαν χώρε οικονομική εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει χώρο για την ανάπτυξη των πολιτικών στι χώρε αυτέ. Επιπλέον είναι ελεύθερε συμφωνίε εμπορίου αυτέ μεταξύ ανισότιμων εταίρων που δεν είναι ισότιμοι. Για το δικό μας λοιπόν συμφέρον και το δικό μας όφελος. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σχεδιάσει ε, πολιτικές και θα επετύχει και τους στόχους της χιλιετία αν εμπόριο απονομεύει τους στόχους που προανέφερα. The floor is now for Mr. Philip Kasmarek. Και τώρα ο κύριος Φιλίπ Κάσμαρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε εδώ για την αναπτυξιακή βοήθεια και όχι μόνο για το πώς τίθεται σε κίνδυνο το ποσοστό του 0,5% αλλά και κάποιοι επιμέρους στόχοι, πολύ βασικοί, το 35% κάποιων χωρών το οποίο διακυβεύεται. Ακόμα και τα κράτη-μέλη που έχουν την απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη τελικά έχουν κίνητρα για να επιδιώξουν τους μερικούς αυτούς στόχους. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή δεν μπορούσε να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη για να καταφέρουμε εδώ κάτι καλύτερο. Ευχαριστούμε ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ. Επίτροπε, να σας συγχαρώ για τις απαντήσεις σας ως τώρα. Ε, ιδιαίτερως με ενδιαφέρουν τα, δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Τι θα κάνετε για να προστατεύσετε τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, ανδρών και γυναικών στον αναπτυσσόμενο κόσμο που συνεχώ δέχονται επιθέσει και είναι θύματα καταπίεση. Τι θα κάνετε για να προστατεύσετε τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίω τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά του δικαιώματα. Ευχαριστώ. Mr. Charles has the floor. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το τελευταίο μου ερώτημα αφορά την επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη και την οικονομική βοήθεια. Κύριε Επίτροπε, θεωρείτε ότι η επιστημονική αυτή βάση είναι αρκετή. Ήθελα να τις εξηγήσεις σας. Κύριε De το λόγο. Για πέντε λεπτά. Merci, Madame la Présidente. C'est vraiment un rythme très soutenu. Mais oui, c'est bien pour Είναι εξαντλητικό ο ρυθμό, κυρία Πρόεδρε. Ανελέητο, ναι, ναι. Κυρία Σαργεντίνη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για συμφωνή σε ελευθέρου εμπορίο. Δεν συμφωνώ. Ξέρετε γιατί έχουμε τέτοιες συμφωνίες προτιμησιακές. Έχουν προηγηθεί συμφωνίες που μας φέρνουν σε σύγκρουση με τις υποχρέωσεις μας προς τον ΠΟΕ και την ΤΟΧΑ. Επομένως είναι σημαντικό και για τις βιομηχανικές αλλά και τις απτυσσόμενες χώρες να είμαστε σύντονοι με τους κανόνες του ΠΟΕ. Δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου. Σα λέω απλώ πώς το σκέφτομαι. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτές οι συμφωνίε είναι μια δίκαιη πρόταση προς τις χώρε ΑΚΕ, προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κάποιε χώρε βέβαια χρειάζονται κάποια προσαρμογή, χρειάζονται και αυτές τις ενδιάμεσες συμφωνίε. που δεν έχονται σύγκρουση με τον ΠΟΕ. Και έτσι εξυπηρετείται και η περιφερειακή συνεργασία. Κύριε Κάτσμαρικ, ελπίζω σωστά προφέρω το όνομά σας. Όντως, κάποια κράτη-μέλη δεν πρόκειται να τηρήσουν τις ε, δεσμεύσεις τους ε, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο τα κάνει η Κομισιόν και το ίδιο το Κοινοβούλιο θα πρέπει κάτι να κάνει. Γιατί και εσείς οι ίδιοι, εδώ εκπροσωπείστε, εσείς εκπροσωπείτε κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις. Επομένως, είναι το σωστό μέρος εδώ να συζητηθεί αυτό το πρόβλημα. Και επίσης είναι λάθος το να μην τηρεί κανείς τα επισχυμένα και πολλά περισσότερα θα πρέπει να κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Κύριε Κάσμαν. Ξέρω το πρόβλημα. Ε, στον Μπουρούντι είχαμε επίσης κάποια θέματα σχετικά με αυτό και παρενέβην για λογαριασμό της ε, χώρας μου γιατί ακόμα τότε ήμουν υπέξ τώρα έχουμε και καινούργιες, ε, καινούργια θέματα σχετικά στην Ρουάντα και εκεί έχουμε νομοθεσία νέα που συζητείται στο Κοινοβούλιο. Έχουμε θέματα σχετικά με φυλακισμένους και συνέταξα μια επιστολή προς τον Γιώργο Καγάμι, τον πρόεδρο της Ρουάντας. ούτω ώστε να παρέμβει και να υπάρξει διορθωτική κίνηση μέσω της νομοθεσίας και να προκύψουν κάποια αποτελέσματα. Αυτό αφορά βέβαια και τα δικαιώματα, τα σχετικά με την ε, αναπαραγωγή, τα γεννητήσια δικαιώματα και αφορά επίσης ε, κάποιες γυναίκες ε, που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σε κάποιες χώρες τώρα όσον αφορά την επιστημονική βάση, όσον αφορά την πολιτική της ανάπτυξης, ε, μας αρκεί. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια τέτοια ε, βάση, βάση επιστημονική. Ε, και πώς να σας το πω, δεν ξέρω, ε, δεν είμαι τόσο σίγουρος για το ότι λαμβάνεται γενικότερα σε όλο τον κόσμο υπόψη το τι επιστημονική τεκμηρίωση υπάρχει. Γι' αυτό και εμείς να λάβουμε την πρωτοβουλία να ζητήσουμε να γίνει μια εξαντλητική μελέτη για τους λόγους βάσει των οποίων έχουμε κακή διακυβέρνηση σε τόσες αναπτυσσόμενες χώρε. Βέβαια αυτό ε, όπως ξέρετε έτσι κι αλλιώς ισχύει εδώ και πολύ καιρό. πάντοτε υπάρχει καθυστέρηση δηλαδή του, του τι, τι πολιτική ασκείται σχέση με το τι έχει εξευρεθεί από τους επιστήμονες. Τώρα προχωρούμε στον 8ο γύρο ερωταπαντήσεων. Εύα Ζανίτσκι. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στα πλαίσια τη διεθνού ε, συνεργασία και οι τοπικοί φορεί, όπω μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι, φορεί αποκεντρωμένε, οι αποκεντρωμένες, τοπική φορείς οι διεθνεί εκπρόσωποι, θα είναι μια ανεκτήμητη συνεισφορά χάρη στι ιδιαίτερε γνώσει του και το απαιτητικό του έργο. Εσεί, ω επίτροπο, πώ σκοπεύετε να ε, έρθετε σε επαφή με αυτού του παράγοντε και να διαλέξετε του πλέον κατάλληλου που θα προσφέρουν και στο δικό σα έργο. Και έπειτα για την απομάκρυνση των ελευθερομεταναστών από την Ιταλική κυβέρνηση. Είναι κάτι πολύ οδυνηρό το οποίο θα πρέπει να αναλύσουμε ει βάθο. Όμω η Ιταλική κυβέρνηση δεν μπορεί να επομίζεται την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Πρέπει να το κάνει αυτό όλη η Ευρώπη και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό σε μια άλλη ευκαιρία ω συζήτηση. Thank you. Mr. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πατρίς Τυρολιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να θέσω το, θέμα της, ε, το, πρωτα, το ζωτικό θέμα τη συνεργασία με τι περιφερειακέ περιοχέ και τι χώρε ΑΚΕΠ. Εάν δούμε τι συμβαίνει στην Αφρική, ε, έχουμε καταφέρει εκεί να αναπτύξουμε τεχνογνωσία σε πολλού σημαντικού τομεί ιδιαίτερου ενδιαφέροντο. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητε συνεργασία με τι ομάδε των χωρών τη Αφρική, αλλά μην ξεχνάμε και την περίπτωση του Καριφόρουμ, όπου βλέπουμε ότι με μεγάλη συνοχή καταφέραμε μια καλή συνεργασία στη ζώνη τη Καραϊβική ε, και για τι χώρε του ΑΚΕΠ αυτό και για την περιοχή του Ειρηνικού. Το Ατλαντικού, μάλλον, συγγνώμη. Οπότε, το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τους πόρους ε, του ΦΕΝΤΕΡ και του ΦΕΝΤ, πώς θα ε, βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ ομάδων χωρών και των χωρών ΑΚΕΠ και τι θα γίνει με τη συνεργασία Βορρά-Νότου σε αυτό το πλαίσιο. Με συγχωρείτε, αλλά έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Το χρόνο έχει ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι που εν μέρει απαντήθηκε από τον Επίτροπο στο οποίο ήθελα να επανέλθω. Το θέμα της ιδιοκτησίας στην χώρα μου τον 19ο αιώνα, τα μέσα και στα τέλη του 19ου αιώνα, είχαμε καταστατικούς λοιμούς, οι οποίοι αποδεκάτησαν τον πληθυσμό της Ιρλανδίας. Το μέρος του πληθυσμού που ανέκαμψε γρήγορα ήταν αυτό το οποίο κατήχε μικρά κομμάτια γης. Έτσι ξεκίνησε βεβαίως και η διέρεση του νησιού μας, αλλά δούλεψε σε εκείνη την περίπτωση. Ποιο θα είναι λοιπόν το έργο της Επιτροπής αυτής. Πρέπει να σταματήσει να μιλάει θεωρητικά για το θέμα αυτό και να αρχίσει να το υλοποιεί, να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους μικροκεφάλαιο, τα δικά, τις δικές τους μικροπεριουσίες και να έχουν κάτι στο οποίο να βασιστούν. Να τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή και να ποιος είναι ένας στόχος που μπορείτε να περιλάβετε στις προτεραιότητές σας. Ευχαριστούμε κυρία Κατού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αναφέρατε στην δήλωσή σας τους υψηλούς αριθμούς των εργαζομένων που έχουν χάσει τη ζωή τους ε, δουλεύοντας σε δυσμενείς συνθήκες Και τα φαινόμενα αυτά αυξάνονται τον τελευταίο καιρό. Τι θα κάνετε λοιπόν για να βεβαιωθείτε για το σεβασμό των διεθνών ε, προτύπων και προδιαγραφών, τον νόμο, ε, το δίκαιο και την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στον χώρο δικαίου, πώ θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και πώ νομίζετε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε το μηχανισμό για τον έλεγχο της κατεύθυνσης των ε, κονδυλίων. Ένα δις δαπανίσαμε, ένα δις ευρώ δαπανίσαμε πέρσι για τους γεωργούς στην Αφρική, αλλά δεν έχουμε καμία γνώση για το πώς δαπανήθηκαν τα ποσά αυτά. Ευχαριστούμε κύριο Κάσμαρεκ. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. σε κάποιες χώρες δεν υπάρχουν θεσμικές υποδομές για την αναπτυξιακή πολιτική. Σκεφτείτε την νομοθεσία, τα εκτελεστικά όργανα, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ε, επίτροπε, δεν θα πρέπει να εμφανιστούν οι χώρες αυτές ώστε να βελτιωθούν ως ε, προς τη θεσμική τους ε, οικοδόμηση, κάτι που θα τους επιτρέψει να γίνουν και καλοί δέκτες της ευρωπαϊκής βοήθειας, της αναπτυξιακής βοήθειας. Κύριε Επίτροπε, έχετε 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Πόσο έχω? 6 λεπτά ολόκληρα και 15 δεύτερα. Ευχαριστώ. Για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις πρέπει να πω ότι είναι ένας απαραίτητος κρίκος ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Διότι πολύ συχνά δεν υπάρχει κράτος ε, συνήθως επιτόπου όταν θέλουμε ανθρωπιστική βοήθεια για να διοχετευτεί αυτή στους αποδέκτες της. Και επιπλέον, όταν υπάρχει κράτος είναι μονοκομματικό, πράγμα που τους καθιστά ακατάλληλους να δράσουν σε μια συγκεκριμένη φάση και στην υπόλοιπη αναπτυξιακή συνεργασία έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν εκατομμύρια κάθε χρόνο, 120 περίπου το χρόνο, 220 συγγνώμη, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες υποβολές αιτήσεων για projects και είναι τρομακτική δουλειά να επιλέξει κανείς. Και πολύ συχνά διαπιστώνω ότι είναι σε πολύ μικρή κλίμακα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε μαζί με όλη αυτή την κοινότητα τον ΜΚΟ πώς θα συντονιστεί αυτό το έργο και το κόστος και πώς θα, κρατηθεί, θα συγκρατηθεί κάπως το κόστος σε συγκεκριμένα πλαίσια, γιατί έχω την εντύπωση ότι σήμερα δεν ισχύει ακριβώς κάτι τέτοιο. Κύριε Τυρολιά, σε ό,τι αφορά τις ε, άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, τις ΡΟΥΙΠ όπως τις ονομάζεται στα γαλλικά, αυτό δεν είναι θέμα του ε, Επιτρόπου Αναπτυξιακής Συνεργασίας, αλλά σε μερικές περιπτώσεις στα γαλλικά είναι dom-tom, δηλαδή ε, απομακρυσμένες περιφέρειες και νομή ε, αλλά έχουν υπερπόντια διαμερίσματα, αλλά έχουν ε, γεωγραφική συνάφεια είναι δύσκολες οι καταστάσεις και πολλές φορές κλιματικές αλλαγές και είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε. Και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΦΕΔ και ΦΕΝΤΕΡ μπορούν να συνεργαστούν για τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες. Κύριε Μίτσελ, για την ιδιοκτησία γης είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι και καθόλου εύκολο, ξέρετε. Έχουμε δει επανειλημμένα απόπειρες να ε, γίνει αναδασμός για παράδειγμα και στο Ζιμπάμπουε αποτέλεσμα ήταν όλεφρος. Και ένα βήμα και πολύ σημαντικό θα ήταν να γνωριστούν τα δικαιώματα ε, τα οποία ήδη είναι κατοχυρωμένα και εκτιμένα δικαιώματα όπου ο κόσμος ε, κατέχει τη γη, αλλά δεν τους αναγνωρίζουν το δικαίωμά τους, τους τίτλους ε, επίσημα. Αυτή τη στιγμή αναγνωριστούν οι τίτλοι ιδιοκτησία, τότε μπορεί αυτό να θεωρηθεί το ενεργητικό τους, ας πούμε, που του δίνουν τη δυνατότητα να δανειστούν κιόλα και να ξεκινήσουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία ενεργητικού αυτά. Οπότε, ακριβώς είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι ιδιοκτήτη της γης του και να έχει και αυτάρκεια. Αλλά επαναλαμβάνω, από πολιτική απόψεω δεν είναι εύκολο καθόλου. Και εδώ επανέρχομαι σε μία ερώτηση του κυρίου Γκέρενς ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη υποστημονική πληροφόρηση και βάση για το πώς θα το κάνουμε αυτά με τρόπο δίκαιο. Γιατί ακόμα και στην Ευρώπη έχουμε δει τέτοια φαινόμενα, ξέρετε. Ε, τα δικαιώματα ιδιοκτησία δεν είναι εύκολα. Αν χρειάζεται να μοιραστεί η γη, αυτό το έχουμε δει, ας πούμε, μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου σε κάποιες χώρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθοριστούν αυτά και ακόμα πιο δύσκολο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά είναι και αναγκαιότητα, αν θέλουμε, να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα κονδύλια που φτάνουν στον κόσμο. Κυρία Κρέτσου, ε, το ανθρωπιστικό δίκαιο. Είναι απορίας άξιο που πέθαναν 122 εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα. Και το μόνο αντίδοτο που θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς είναι να τονίζουμε πάρα πολύ την ανεξαρτησία και την ε, αμεροληψία όλων αυτών των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή ε, μπουν σε μια πολιτική στρατηγική αυτή και εμπλακούν, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η θέση τους και ευάλωτη. Και θα πρέπει να τους προστατεύουμε. Στον Ταρφούρ, για παράδειγμα, είχαμε δυστυχήματα, πολλά είναι προφανές ότι αν είχαμε εκεί στρατεύματα θα βοηθούσε την κατάσταση αυτό και θα ήταν πιο αποτελεσματικό και θα είχαν αποφευχθεί. Έχουμε λοιπόν εκεί μια διάδραση. Από τη μια χρειάζεται αρκετή προστασία, αλλά να είναι τελείω ανεξάρτητη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεξάρτητοι, κινδυνεύουν. Και ακριβώς το ίδια ισχύουν και με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό αυτή τη στιγμή δεν είναι τελείω ανεξάρτητοι, μπαίνουν σε μπελάδε και οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν μπορώ ακόμα να απαντήσω την ερώτηση του κυρίου Κάσμαρεκ. Ναι, εντάξει. Απαντήστε. Τη. Σε πολλά κράτη-μέλη το θέμα είναι ότι λείπει η θεσμική υποδομή που είναι απαραίτητη για την αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό ισχύει και σε εθνικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ περίπλοκα πράγματα. Και νομίζω θα έχει μεγαλύτερο νόημα να βοηθήσουμε τα νέα κράτη-μέλη να φτιάξουν τέτοιες υποδομές. Αλλά αυτές οι υποδομές θα πρέπει να γίνουν με τρόπο ώστε να μην γίνει εις βάρος των όσων συμβαίνουν στα διάφορα ήδη υπάρχοντα κράτη-μέλη. Αλλιώς θα ήταν μια τρύπα στο νερό. Καλύτερα να διοχετεύσουμε προς την Ευρώπη αυτή την προσπάθεια που να είναι πρωταγωνιστή σε εκείνη, για να μην έχουμε επικαλύψεις. Thank you. We will now start the last question round for the members of this committee. Τώρα ο τελευταίος γύρος ερωτήσεων για τα μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Μιγγέλ Μαρτίνες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση με την Αφρικανική Ένωση για την επομένη συνάντηση κορυφή που θα γίνει περίπου σε ένα χρόνο, συνάντηση κορυφή Αφρική-Ευρώπη. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε τα θέματα της χρηματοδότησης όσον αφορά την κοινή στρατηγική. Ε, τώρα η χρηματοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Κάτι το οποίο ξεκίνησε από την προηγουμένη συνάντηση κορυφή. Τέλος δε, στα γαλλικά αναφέρατε κύριε Επίτροπε, αυτό το οποίο είπε ο προκάτοχός σας. Αν δεν το κάνετε από ελεγγύη, κάντε το από συμφέρον. Εγώ λέω κάντε το από για το ότι το, το, επιτάσσει η λογική. επόμενος. Ναι, Είπατε στο βελγικό τύπο ότι θέλετε να επαναφέρετε τη θεσμική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα τονίσατε την έλλειψη πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το Συμβούλιο και την επικρίνατε. Εσείς πώς φαντάζεστε τη μελλοντική θεσμική ισορροπία στον τομέα της αρμοδιότητάς σας και τι επιπτώσεις θα έχει η δική σας δέσμευση ε, στους όρους και σχέσεις συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το λόγο έχει η κυρία Ντεκάιζερ. Κύριε Ντεγκούχτ, η ειλικρίνειά σας είναι πραγματικά μυθική. Λέτε δυνατά αυτό που κάποιοι το σκέφτονται μόνο χαμηλόφωνα. Λέτε κάτι λοιπόν που για την Επιτροπή μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες, καθώς και διπλωματικά το ίδιο για τη διακυβέρνηση κάποιων χωρών που αναφέρατε. Τι εγγύησεις μπορείτε εσείς να μας δώσετε ότι δεν θα υπάρξουν αυτές οι ε, ανεξέλεγκτες διπλωματικές συνέπειες που φοβόμαστε, αυτός ο εκτροχιασμός που μπορεί να προκύψει. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Αξέρα, ο κύριος μάλλον. Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο ο μιλητής. Ευχαριστούμε. Είπατε ότι μια ψηφοτεραιότητας είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση στις πιο φτωχές χώρες. Ωραία αυτά τα λόγια, αλλά πέστε μας τι συγκεκριμένα μέτρα θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σκοπό. Και πέστε μας κατά πόσον πρόκειται να διατεθεί κάποιο συγκεκριμένο κονδύλιο πάλι για αυτό το λόγο. Πρόεδρος. Έχουμε χρόνο, οπότε μπορεί να υποβληθεί ακόμα μια ερώτηση. Θα προέρχεται. Κυρία Ελένη Θεοχάρους, παρακαλώ. Okay. I'm sorry. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο κύριος Μίτσελ μας είπε προηγουμένως ότι προβλήματα ιδιοκτησίας οδήγησαν σε τελική ανάλυση την Ιρλανδία στη διέρεση. Εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στη δικιά μου τη χώρα η βίαιη ε διέρεση έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην ακτιμοσύνη και στην προσφυγοποίηση και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Ε, στην ερώτηση μου τώρα προς τον κύριο Επίτροπο, είναι γνωστό ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες απομιζούν το επιστημονικό δυναμικό αλλά και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό επαγγελματίες όπως είναι οι νοσηλευτές, οι ΜΕΣ, οι τεχνικοί από τις αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως από την Αφρική. Και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας που προάγει την υποανάπτυξη. Thank you. Ολοκληρώσαμε το κύριο ερωτήσεων για τον Επίτροπο. Αλλά θα θέσω και εγώ ένα ερώτημα προς τον κύριο Δεκούχτ. Ακούσαμε τους πάντες να λένε ότι ανησυχούν ιδιαίτερα με την κατάσταση. Γιατί υπάρχει χάσμα μεταξύ αναγκών και πόρων. Είναι πάρα πολύ βαριές οι ευθύνες που πρέπει να αναλάβουμε εφ' Θα σας ρωτήσω λοιπόν ποιες είναι οι προθέσεις σας έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών και τις δικούς τους πόρους. Τι θα κάνετε εσείς για να βοηθήσετε τις αναπτυσσόμενες χώρες να διατηρήσουν αυτούς τους πόρους που ενδεχομένως έχουν στην κατοχή τους και να βελτιώσουν και το φορολογικό τους εισόδημα. Κύριε Επίτροπε, Έχετε 6 λεπτά αυτή τη φορά και 15 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Μαρτίνες. Ε, Μαρτίνες. ως ε, Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής προετοιμάζεται εντατικά στο Συμβούλιο. Ήδη στις 15 Οκτωβρίου θα υπάρξει και Τρόικα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αφρικανικής Ένωσης που αν δεν απατώμε θα γίνει στην Αντίσα Μπέμπα, έτσι. Και στο μεταξύ, σε επίπεδο διοίκησης ε, και υπηρεσιακών επαλλήλων ε, προετοιμάζεται ε, είναι 8 οι τομεί και καταγράφεται η πρόοδος που έχει γίνει σε αυτού του τομεί συνεργασίας. αυτό το καιρό. Τώρα, το θέμα της θεσμικής ισορροπίας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε θεσμικό όργανο να διαδραματίζει το ρόλο που του αναλογεί ε, στο θεσμικό οικοδόμημα. Και ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακριβώ να κάνει τι προτάσει. Έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία, όπω λέγεται. Και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει το δικαίωμα πρωτοβουλία και μην αφήσει να τη το ψαλιδίσουν. Ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σε σημαντικό βαθμό συνεργασία με το Συμβούλιο να είναι τα δύο σώματα του κοινοβουλευτικού συστήματος. Και είναι σημαντικό ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μπάλιν, γιατί εξορισμού είναι ε, τα δύο θεσμικά όργανα που ε, καλούνται να υλοποιήσουν και να υπερασπιστούν το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί από τη συνθήκη. Και δεν θα πρέπει να ψάχνουν για εναλλακτικέ λύσεις έτσι κάπως Κυρία Ντεκάιζερ, με ικανοποιεί ιδιαίτερα το ερώτημά σας, διότι λέτε ότι εκφράζω δυνατά αυτό που άλλοι το σκέφτονται μόνο χαμηλόφωνα, αλλά φοβάμαι και τις διπλωματικές συνέπειες. Αλήθεια είναι και αυτό, αλλά επίσης αλήθεια είναι ότι όταν κανείς ακριβώς δεν φοβάται να πει την αλήθεια ανοιχτά, κάποιοι αντιδρούν έντονα σε αυτή την αλήθεια. Όταν δούλεψα ως Υπουργός Εξωτερικών για πέντε χρόνια, μου συνέβη αυτό. Και με τον πρόεδρο Καμπίλα συγκεκριμένα. Και πριν πήγε, πάω στην Κινσάσα, είχα πει ότι θα πρέπει να μιλήσουμε κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο στα μάτια για να βγει άκρη. Είναι λοιπόν σημαντικό και το στοιχείο της ανθρώπινης επαφής αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Εξέλα, Όντως υπάρχουν συμπληρωματικά μέτρα και μέσα για την αντιμετώπιση κατεπηγόντων προβλημάτων ε, και μετά την κρίση. Ε, είναι το μέσο, μέσο flex, ε, αν δεν απατώμε, 500 εκατομμύρια για το 2009-2010 και ε, τραβηχτικά δικαιώματα που απορρέουν από τη συμφωνία του Glen Eagles. Αλλά επίσης είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε ότι στα χρηματοοικονομικά μέσα είναι πολύ λίγα αυτά που κάνουμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, τα κανονικά ε, κράτη-μέλη να λειτουργούν και κανονικά εντός εισαγωγικών ε, στη σημερινή κατάσταση της οικονομικής κρίσης που ζούμε. Και έρχομαι στην ερώτηση της Προέδρου αν δούμε τι γίνεται με τις χρηματικές ροές, την αναπτυξιακή συνεργασία και τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι προφανές ότι έχουμε δύο ρεύματα. Την αναπτυξιακή βοήθεια και ε, επίσης κάποια άλλα εμβάσματα που είναι τα διπλάσια από την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά θα πρέπει για να απτυχθεί μια χώρα να έχει και εσωτερική ανάπτυξη και φορολογική δυνατότητα ε, και ε, φοροεισπρακτική δυνατότητα. Ε, αυτό είναι ένα έδαφος που πρέπει να διερευθυνθεί. Να αναπτύξουν αυτή τη δυνατότητα πρώτον οι αναπτυσσόμενες χώρες και να το πω κάπως μετριοπαθώς. Η διαφθορά που συνδέεται με όλα αυτά να Πώ ψάχνω να βρω την κατάλληλη λέξη, να αγωγηθεί κάπως, να τηρηθεί με εντό ορίων. Και θα πρέπει να επιβάλλονται και φόροι. Και στην Ευρώπη ε, πάντα οι φόροι επιβάλλονται παραδοσιακά στην πηγή θα μπορούσε να γίνει αυτό και στην Αφρική με βάση την παραγωγή και να γίνεται φορολόγηση στην πηγή. Έτσι παθαίνει μια χώρα να μαζεύει φόρους. Έτσι αναπτύσσεται. Επίσης, και θα ήθελα ε, και είμαι στη διάθεσή σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, να το εξτάσουμε αυτό. Για την Κύπρο, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αποφανθώ. Δεν νομίζω να είστε αρμοδιότητες. Μιλήσατε κι εσείς για τη διαρροή εγκεφάλων. Υπάρχει πρόβλημα σίγουρα και το θέμα είναι ακριβώ η συνέπεια και η συνέχεια και η συνοχή στην αναπτυξιακή μα συνεργασία. Δεν έχει νόημα από τη μια να δίνουμε χρήματα για την ανάπτυξη των χωρών αυτών και την κατάρτιση κάποιων προσώπων, στη συνέχεια να του φέρνουμε αυτού στην Ευρώπη επειδή έχουμε έλλειψη στην Ευρώπη ε, τέτοιων ε, μυαλών. Σίγουρα εδώ χρειάζεται συνέπεια και συνοχή στην πολιτική μας. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους. Πριν πριν όμως κηρύξω τη λήξη της συζήτησης αυτής, θα δώσω και πάλι το λόγο στον Επίτροπο, εφόσον το επιθυμεί, για κάποιες καταληκτικές πρατηρήσεις. Έχετε περίπου τρία λεπτά. Euh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προσπάθησα στον χρόνο αυτό που μου δώσατε για τις απαντήσεις να καλύψω μέσα σε μια μισή ώρα που είναι αδύνατον όλα τα θέματα όλα αυτά που σας απασχολούν. Οπότε θα ήθελα να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας τους αμέσως επόμενους μήνες όταν θεωρείτε ότι ε, χρειάζεται να έρθω στην Επιτροπή σας να συμμετάσχω στις εργασίες σας. Πρώτα πρώτα. Είχαμε το θέμα του συναδέλφου μου, ο οποίος θεώρησε ε, ότι καλό να ρωτήσει αν πρόκειται να δουλέψουν με σοβαρότητα. Βεβαίω και αυτό θα κάνω. Το έκανα αυτό και στο παρελθόν. Όποτε είχα κάποιο πολιτικό αξίωμα και γι' αυτό και πιστεύω αυτούς ε, μέσω επόμενους ε, μήνες ε, να εργαστώ πάνω σε αυτά τα θέματα και να βοηθήσω στην άσκηση αυτής της πολιτικής εκ τη της ε, ε, Κομισιόν για την αναπτυξιακή συνεργασία. Θα είναι βεβαίω ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια και της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την χρηματοδότηση τα θέματα τα σε σχέση με το κλίμα, με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε να κάνουμε πολύ σοβαρή χρηματοδότηση, να βοηθήσουμε με βιώσιμο τρόπο τις ε, χώρες που εμπλέκονται. μια που υπάρχουν κάποιοι φόβοι ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης ε, όπως ήταν αυτοί πριν την οικονομική κρίση και φοβόμαστε ότι αυτό επομένω θα, θίξει, θα πλήξει πάρα πολύ τι αναπτυσσόμενε χώρες. Επομένω, έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ προκλήσει μπροστά μας. Αυτό θα απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά επομένως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμένα συγκεκριμένα του αμέσω επόμενου μήνε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε υποψήφιο Επιτροπέ για τις απαντήσεις σας. Θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξη, μια που ποτέ μέχρι τώρα δεν ε, είχαμε τέτοιες ε, προκλήσεις. Έχουμε αυτούς τους στόχους, ε, τους δύο βαθμούς, ε, σαν στόχο. Ε, οπότε, με μεγάλη μας χαρά, συμφωνούμε με την ιδέα σας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν βεβαίως είναι θετική η γνωμοδότηση, βλέπουμε μας μεγάλη μας χαρά ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ έντονη συνεργασία τα μέσα επόμενα χρόνια. Εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την συνάντησή μας και σας ευχαριστούμε που τηρήσατε όσο επιτοπλίστων τα χρονικά όρια. Θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα γιατί έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Και ήδη ε, έχουμε μείνει πίσω. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους.